Good morning, ladies and gentlemen. Let start. Uh, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε τη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ήτρε. We go to the uh, next point. Θα περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του, ε, της χειμερινής δέσμης μέτρων. Εισηγητής είναι ο Κλοντ Τούρμες. Στις 30 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο καθαρής ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους. το οποίο συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ενεργειακή ε, απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, ασφάλεια εφοδιασμού, ασφάλεια ε, της αγοράς και κανόνες διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση. Και συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες διακυβέρνησης εδώ. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συνεχίσουμε την συζήτηση για το χειμερινό αυτοπακέτο και θα συζητήσουμε δύο θέματα. Καταρχάς, τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Θα καλέσω επίσης και την κυρία Ριβαζή. Α, δεν θα έρθει, δεν θα έρθει. Η κυρία Ριβαζή είναι η συγκήτρια της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης διότι όπως γνωρίζουμε όλοι καλά, η Ενεργειακή Ένωση συμπεριλαμβάνει και περιβαλλοντικά ζητήματα, εκτός από την ενεργειακή απόδοση που είναι δική μας αρμοδιότητα. Όμως, ε, λόγω της ε, περιβαλλοντικής διάστασης συμπεριλαμβάνεται και η Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ. Επίσης θα συζητήσουμε την οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης η οποία φυσικά είναι μία οδηγία που αφορά μέσα την Επιτροπή μας. Η συγητής είναι ο Άνταμ Γκίρεκ και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εδώ όλους τους συγητές και τους σκιώδεις. Θα θέλατε να πείτε κάτι, αγαπητοί συνάδελφε. Θα αρχίσουμε με τη διακυβέρνηση. Ναι. Το λέω πάντα πως όλοι οι συγητές που ασχολούνται με τα θέματα του χειμερινού πακέτου θα ήταν καλό να είναι μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτό δείχνει μεγάλη υπευθυνότητα. Χρειάζεται συντονισμός, ξέρετε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται και πού βρίσκονται οι άλλες προτάσεις. Αρχίζουμε λοιπόν με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Συνάδελφε Τούρμες, έχετε το λόγο. Πόσο χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε? Πέντε λεπτά. Όπως πάντα. Το 2016 ήταν η θερμότερη χρονιά από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις. Και διαβάσαμε ότι και ο πάγος της Αρκτικής και της Ανταρκτικής βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 35 ετών. Γιατί το λέω όμως αυτό. Διότι υπάρχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται επίγουσα δράση. Το καλό είναι ότι υπάρχουν και λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε καταφέρει τα τελευταία 15 χρόνια, ειδικά εμείς εδώ στην Επιτροπή. Θέσαμε τις βάσεις για να γίνουν φθηνότερες οι λύσεις, δηλαδή η αιωλική ενέργεια, η ε, η ηλιακή ενέργεια είναι φθηνότερε από ποτέ, είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Γνωρίζουμε επίσης πώς να κατασκευάζουμε ε, σπίτια ουδέτερης ενέργειας ή και θετικής ενέργειας. Μπορούμε να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας και να τα μετατρέψουμε έτσι ώστε να είναι πιο ε, μονομένα. Αυτή η πρόοδος έχει συνοδευτεί και από νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για εξαγωγές. Έχει επίσης συμπεριλάβει πιο καθαρό αέρα. Έχουμε ωφέλη. Γι' αυτό θεωρώ πως τον κανονισμό περί διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης πρέπει να δώσουμε έμφαση στο πώς αυτή η μετάφαση που χρειάζεται, που είναι απαραίτητη, θα γίνει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος επενδύσεις που γίνονται, είτε είναι σε ανανεώσιμε, είτε σε ηλεκτρική κινητικότητα, είτε σε ανανέωση κατοικιών, πρέπει να γίνονται με χαμηλό κόστος. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι γιατί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ε, στοιχείων στην Πολωνία ε, ε, παράγει ενέργεια που κοστίζει 95 ευρώ την, ε, τη μεγαβατόρα και στην ε, Δανία 55. Γιατί στην ε, Ρουμανία ο επενδυτής ε, πληρώνει περισσότερα για μια επένδυση στη Ρουμανία από ότι ένας Γερμανός επενδυτής στη Ρουμανία. Υπάρχει λοιπόν θέμα και πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα και εννοώ το πώς αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο οι επενδυτές. Γι' αυτό ο κανονισμός ε, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης μπορεί να έχει ε, πολύ σημαντικές ε, θετικές συνέπειες. Καταρχάς χρειάζεται σαφήνεια για το τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε. Είναι λοιπόν σημαντικό η Επιτροπή αυτή να έχει πολύ σαφή, λεπτομερή σχέδια για το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2050 πρέπει να μειώσουμε τον ε, στόχο μας στο μηδέν. Και η τάση που υπάρχει γνωρίζετε είναι να αποφεύγουμε ε, την πραγματικότητα. Να λέμε εντάξει, αργότερα, προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Για να περάσουμε στα, από το 27% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 100% με, ε, στα επόμενα 20 χρόνια, μπορείτε να καταλάβετε ότι ε, θα χρειαστούν πολλά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν γίνεται αν συνεχίσουμε έτσι. Ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί το κόστος ε, πέρα από τις επενδύσεις είναι και να ε, αυξηθεί η αποδοτικότητα. Αυτό συνεπάγεται καλή συνεργασία. Υπάρχει και μία σχετική μελέτη που αφορά το κόστος της μη συνεργασίας ή της κακής συνεργασίας. Μετά, στην Ευρώπη ζούμε δύσκολες εποχές και γι' αυτό χρειάζονται έργα μεγάλης ε, ορατότητας. Χρειάζεται ας πούμε να γίνουν μεγάλα έργα στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική, ανεμογεννήτριες, συλλογική δράση στην Κεντρική Ευρώπη έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ηλεκτρική κινητικότητα. Και για να μην αναφερθούμε στους ε, συναδέλφους μας από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ε, ηλιακής ενέργειας. Υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται με το οικονομικό κόστος των επενδύσεων στις ανανεώσιμες, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Οι κυβερνήσεις δεν είναι μόνοι, μόνες τους. Οι πολίτες δεν είναι ε, μόνοι τους αυτό. Χρειάζεται μία συνεργασία, μία συλλογική προσπάθεια, διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτή. Μία πόλη, ας πούμε, δεν μπορεί να ε, εφαρμόσει Λύσει χωρί τη συνεργασία τη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να επιτύχει στόχου χωρί βοήθεια και αντίστοιχα η κυβέρνηση χωρί τι προσπάθειε των πολιτών μια πόλη δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Χρειάζεται λοιπόν συμπερίληψη όλων των ε, ομάδων σε αυτή τη διαδικασία, από τον πολίτη μέχρι την κυβέρνηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κάριν έχει το λόγο, εκ μέρου του ΕΛΚ θα αντικαταστήσει τον σκιώδη κύριο Χόκμαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Γκούναρ Χόκμαρκ και θα διαβάσω μία δήλωση που προετοίμασε ο συνάδελφος που δεν ήρθε σήμερα. Τώρα θεωρείστε πως είμαι ο Γκούναρ. Θα αρχίσω λέγοντας πως είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να εργαστούμε αποδοτικά και ταχύτατα για αυτό το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Η Ενεργειακή Ένωση και η διακυβέρνησή της είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Πάλι γκούναρη είμαι, ακούστε εσείς. Θα ε, συνεργαστώ λοιπόν με τον ε, εισηγητή κύριο Τούρμες και με τους υπόλοιπους κοιόδης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ε, προβλεψιμότητα και συγκρισιμότητα των αγορών ενέργειας. Ε, ο Γκούναρ επίσης ε, θα κάνει κάποια πρόσθετα σχόλια. Λέει ότι η Ενεργειακή Ένωση καταρχάς είναι ένα από τα σημαντικότερα ε, project της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δεδομένα των γεωπολιτικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια, για να υπάρχει μια λειτουργική αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα χαμηλώσει τις τιμές και θα δώσει ωφέλη στους πολίτες και ε, θα διασφαλίσει ενεργειακή απόδοση, διασυνδέσεις δικτύων και ασφάλεια εφοδιασμού, χρειάζονται συγκεκριμένα συστήματα, μηχανισμοί, κοινό σχεδιασμό, υποβολή εκθέσεων, έλεγχοι, έτσι ώστε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Δεύτερον, με καλό σχεδιασμό ο διοικητικός φόρτος θα μειωθεί σημαντικά. Αυτό θα γίνει ε, εναρμονίζοντας όλες τις ε, σημαντικές υποχρεώσεις σχεδιασμού, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ε, ο σκοπός του συστήματος διακυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζει την συγκρισιμότητα και την προβλεψιμότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας παρά να επιβάλλει πρόσθετα το ε, άχθος ε, και ε, περιττή γραφειοκρατία. Επίσης, αυτό το σύστημα διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να οδεύει προς μια ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας που θα είναι ικανή να αντέξει σε κρίσεις και εξωτερικές πιέσεις. Επίσης, ο σχεδιασμός των υποδομών είναι εξίσου σημαντικός και πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του κυβερνητικού σχεδιασμού γι' αυτό. Ο Γκούναρ επίσης, εγώ δηλαδή, ε, ε, θεωρεί πως πρέπει να βρούμε τρόπους η διακυβέρνηση και η κυβέρνηση να ε, μην επιβαρύνεται τόσο πολύ στην υποβολή εκθέσεων και στους ελέγχους. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε, να εισαγάγουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την, το ένα οικονομικό κόστος. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν μένουμε στάσιμοι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, περάσαν τα δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο μπορώ να διαβάσω και το υπόλοιπο. Ναι, πολύ σύντομα να το κάνετε όμω αυτό. Ναι, αν τα διαβάσω γρήγορα θα θυμώσουν οι διεμηνεί. Τέταρτον, το σύστημα διακυβέρνηση πρέπει να είναι ευέλικτο και να λαμβάνει υπόψη τι αφετηρίε και τι επιθυμίε όλων των κρατών μελών. Και τέλο, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ε, δώσει προβλεψιμότητα στον σχεδιασμό. Και η ε, Ενεργειακή Ένωση έχει στρατηγική σημασία. Πρέπει να είναι δομημένη πάνω σε συνεργασία, σε αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει τον, την αναγκαία υποστήριξη. Σα ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ο Γκούναρ ε, θα χαρεί πολύ να συνεργαστεί με του υπόλοιπου. Η κυρία Γκρίφιν, εξ ονόματο ε, των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία τα είπατε. Συνάδελφοι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κλόντ ε, για ε, την παρέμβασή του. Συμφωνώ απολύτω με τον Κλόντ ότι χρειαζόμαστε υψηλά επίπεδα φιλοδοξία. Οι σοσιαλδημοκράτε εργάζονται ήδη από κοινού με τον Κάρλο Σερίνο, που είναι σκιώδη ε, στην ΕΝΒΗ, και με του συναδέλφου από την Οριζόντια Ομάδα Εργασία, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ισχυρή διασύνδεση μεταξύ όλων των φακέλων αυτού του πακέτου. Επί του περιεχομένου πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε αυτόν τον κανονισμό. Πρώτον, θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για να διευκολύνουμε την ενεργική μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκέντρωση της παραγωγής, ναι, ανάπτυξη των ΑΠΕ, ε, στόχοι ε, ενεργειακής απόδοσης, όλα αυτά δεν είναι δεδομένα και ούτε λιμένα. Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα εργαλεία ένα σημαντικό στοιχείο είναι η χρηματοδότηση. Γι' αυτό θέλω να συνδέσουμε το κανονιστικό πλαίσιο με ευρωπαϊκέ λύσει χρηματοδότηση. Αυτό θα δώσει κίνητα και για τα κράτη-μέλη και για του επενδυτέ επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα διευκολύνει την ικανότητα προγραμματισμού των κρατών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση στους εργαζόμενους στις δεξιότητες. Όμως αυτό ενέχει και ισχυρή δέσμευση από πλευρά μα, απαιτεί τέτοια δέσμευση, σε ό,τι αφορά τους στόχου μεγική απόδοση και τις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για να δώσουμε ασφάλεια στου επενδυτές και βεβαιότητα. Μετά έχουμε και τις, τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές από τον άνθρακα που έχουμε αναλάβει Το 2018 μάλιστα θα έχουμε τους νέους στόχους μέχρι το 2030. Όμως ε, υπάρχει ασυνέπεια εδώ. Θεωρώ ότι θα πρέπει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να διαμορφώσουμε στόχους συγκεκριμένους ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να αυξηθεί το κόστος ε, των εκπομπών. Μετά θα πρέπει να μα απασχολήσει και η μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050. Δεύτερο βασικό στοιχείο θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλο των ε, ενδιαφερμένων μερών. Και τέλο, ε, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και στα εθνικά σχέδια διατάξεις για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή ένδυα. Και κάτι τελευταίο, να ευθυγραμμιστούμε με τους στόχους της COP21, τη διαφάνεια και τη συμπερίληψη των ενδιαφερμένων μερών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ πιο σύντομοι από τον Κούναρ και τον Κρίστιαν. Ο συνάδελφος το Σινόφσκι από τους ε, στρατικούς μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, εκτιμώ ιδιαίτερος το γεγονός ότι ο κύριος Τούρμες μας έστειλε γραπτός τις προτάσεις του για την προσέγγιση της έκθεσης αυτής. Έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για τη συζήτηση. Εκ πρώτης όψεως, εκπλήσωμε που ο Κλοντ αναφέρει τόσο φιλόδοξους στόχους ενεργικής απόδοσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρώτη αύξηση μέχρι το 20 μπορεί να είναι δύσκολη γιατί οι ψηλότεροι στόχοι πάντα είναι πιο δύσκολο να επιτευθούν. Διαβάζοντας κανείς ε, την έκθεση, βλέπουμε ότι επιθυμούμε ε, την ότι χρειάζεται να τα επαναξετάσουμε αυτά σε επιμέρους ε, εκθέσεις. Είναι σημαντικό να υπάρξει όμως και εναρμόνιση μεταξύ των ε, επιμέρους αυτών εκθέσεων. Έχω και μια επιφύλαξη εξαιτίας των οικονομικών ε, διαστάσεων. Ίσως να μην είναι εύκολο να εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά κάψιμα, γιατί με το να συντομεύουμε ε, το προσδόκιμο ζωής αυτών των εγκαταστάσεων, αυτό μπορεί να έχει ε, συνέπειε συνέπειες ε, στους επενδυτές και παρόχους που ε, διασφαλίζουν ένα σταθερό περιβάλλον στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πλουστεύσουμε όντως τις δομές και το περιεχόμενο των εθνικών εγκαταστάσεων και θα πρέπει η έκθεση να απλουστευτεί και να γίνει πιο σύντομη. Θα είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν αυτά τα εθνικά σχέδια μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Και κάτι τελευταίο. Εμέσως θεωρώ ότι παρεμβαίνουμε στο ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών. Αυτό με προβληματίζει. Βάσει τις συνθήκες Λισαβόνα. όλα αυτά υπάρχονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριο Σταμποράνο τώρα από το EFDD. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την ε, εισήγηση του, του ε, υπεύθυνου και

Ο στόχος 27% μέχρι το 2030 και το 30% για την απόδοση είναι φιλόδοξη για να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους του 2050 και για να τηρήσουμε τη Συμφωνία του Παρισιού. Νομίζω πως ε, θα έπρεπε να προχωρήσουμε τουλάχιστον στο 45% για τους ανανεώσιμες και ε, στο 50% για ε, την απόδοση. Επιπλέον θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματική και να μπορούμε να μετρήσουμε τα όσα έχουμε ορίσει όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες ε, οι διστάσεις ε, των κρατών μελών, είτε, θεσμική, είτε, είτε θεσμικές είτε λόγω διαφόρων συμφερόντων, θα είναι καλύτερο να ε, καμφθούν μέσω συγκεκριμένων στόχων. Η εμπειρία αυτό μας διδάσκει. Δεν θα θέλαμε στη διάρκεια των ετών κάποιες χώρες πιο πονηρές να προχωρήσουν σε μια ενεργειακή μετάβαση όπως η Δανία ή η Ισπανία, ενώ άλλες χώρες να μείνουν πίσω όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Ισπανία και να πέσουμε και πάλι στην σκλαβιά την ενεργειακή. Αντί να, εξα... να εξαρτώμαστε από την Μέση Ανατολή, τη Ρωσία ή τη ΣΥΠΑ, να εξαρτώμαστε από τα άλλα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπιστούν τα ε, θετικά ευρωπαϊκά project που θα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε επίπεδο κρατών. Τώρα τα κοινά project έχουν μόνο υποδομέ για, τα... για το φυσικό αέριο, τα, ορυκτά, τα αστεριά καύσιμα και όχι για τις ανανεώσιμες που θα έπρεπε να εντοπιστούν και να χρηματοδοτηθούν τα project αυτά με τα υπάρχοντα μέσα, να είμαστε αξιοπρεπείς και να θεωρήσουμε ότι αυτές οι υποδομές είναι, ότι αυτά τα μάλλον τα έργα είναι υποδομές. Και τέλος για το κόστος και για να συνδεθώ με τα όσα έλεγε και ο συνάδελφος Τούρμες, στην Ευρώπη όχι μόνο υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στην Ιταλία ακόμα και ανάμεσα στις περιφέρειες υπάρχουν διαφορές. Όταν ας πούμε έχουμε κρατικές προμήθειες, ας πούμε για τα φωτοβολταϊκά, όχι μόνο υπάρχουν σημαντικές διαφορές, αλλά και το ακόστη δένονται με τα όσα γίνονταν πριν από χρόνια, όταν όλα αυτά κόστιζαν πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Σαφχάουζερ από το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω και μπορούμε να στηρίξουμε τους φιλόδοξους ε, στόχους ε, και θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω κάτι. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως ε, πατριαρχική δομή και με συγχωρείτε και αυτό που λέω. Είναι σαν να λέμε ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσέχει λίγο τα παιδάκια της που είναι τα κρατημέλη, ε, τα προσέχει από πριν, κατά τη διάρκεια, μετά, να δει αν φέρονται καλά και αν όντω ακολουθούν τους κανόνες και τους στόχους που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη βεβαίω του Κοινοβουλίου και εμείς είμαστε όλοι πέρα αυτών των πολύ φιλόδοξων στόχων. Εγώ είμαι υπέρ μια ε, πολύ περισσότερο φιλελεύθερη ε, πολιτική, λιγότερο πατριάρχική. Δεν θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη είναι παιδιά που πρέπει να του λέμε κάθε φορά τι πρέπει να κάνουν και ότι είναι αρκετά υπεύθυνα από μόνα του, είναι λογικά και ξέρουν κατά κάποιον τρόπο τι πρέπει να κάνουν και πρέπει πάνω απ' όλα να του δώσουμε τα μέσα για να μπορέσουν όντω να πετύχουν ε, του στόχου που θέλουν και τα αποτελέσματά του. Επομένω, η άποψή μου είναι η εξή. Πρώτον, τα χρηματοδοτικά μέσα τι νόημα έχει να δίνουμε στόχους αν δεν δίνουμε τα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτά τα μέσα λοιπόν σήμερα δεν τα έχουν πλέον τα κράτη-μέλη εξαιτία των δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά και επειδή δεν έχουν πλέον την ε, ε, νομισματική του κυριαρχία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα που είχαμε παλιότερα να κόψουμε χρήμα για να κάνουμε επενδύσει στην ενέργεια. Σήμερα λοιπόν αυτά τα μέσα τα αρνείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνει και στόχου που είναι απολύτως ανέφικτοι. Δώστε μα λοιπόν τα χρηματοδοτικά μέσα, α εφαρμόσουμε μία... Ε, στρατηγική που να συνδυάζει την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι θεμελιώδες ε, θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε ακριβώς ε, αυτή τη στάση, τη θέση ε, των κρατομελών, δίνοντάς τους τα χρηματοδοτικά μέσα. Για κάτι τελευταίο κύριε Πρόεδρε, βεβαίως και είμαι υπέρ της ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Πρέπει πρώτα να προωθήσουμε τις οικονομίες ενέργειας, ε, την εξοικονόμηση μάλλον και μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέγει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέλη τώρα. Και ο κύριος Ζαμονάτο, επίσης συζητητής για την καθαρή ενέργεια. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτή τη φάση της συζήτησης ε, πολλά πράγματα έχουν ήδη και εγώ ιδιαίτερα συμφωνώ με τα όσα λέει ο Κλοντ. Εδώ παίρνω το λόγο για να εκφράσω εν γέννη τη στήριξη στην, στον νέο κανονισμό που, υπέβαλε, που παρουσίασε η, η Κομισιόν. Μια λειτουργούσα ενεργειακή ένωση χρειάζεται βεβαίως μια ε, διαφανή και αξιόπιστη διακυβέρνηση και μια προοπτική ε, μακρόχρονη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μου, το κόστο του σχεδιασμού των αναφορών και της παρακολούθησης να, απλοποιηθεί και να ανάγονται όλα αυτά σε ίδια λογική, δημιουργώντας ένα κατάλληλο ε, πλαίσιο για την επίτευξη αυτού των στόχων το 2030 για την ενέργεια και το κλίμα. Όπως συχνά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα κάτι μέλη θα πρέπει να αφήνουν την διεθνική τους ε, ε, ε, στάση όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Θέλω να τονίσω λοιπόν την σημασία των προκλήσεων που έχουμε ενώπιόν μα. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε την επίτευξη ορισμένων στόχων στην απόδοση αλλά και για τι ανανεώσιμε Και είναι σαφέ ότι σε αυτό το πλαίσιο η αξιοπιστία των εθνικών ολοκληρωμένων σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα είναι το βασικό ε, μέσο που έχουμε στη διάθεσή μα για να εξασφαλίσουμε την ε, επίτευξη αυτών των στόχων. Καλό είναι λοιπόν να ε, επιβλέπει η Κομισιόν και να προτείνει μέτρα σε περίπτωση που τα εθνικά πλάνα δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Όμως δεν νομίζω πως αυτό μόνο μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές την απαραίτητη ε, ρυθμιστική ε, βεβαιότητα και σταθερότητα. Είναι ευκαιρία για επενδύσεις και για να γίνουν επενδύσεις πρέπει οι επενδυτές να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Η Ευρώπη λοιπόν για να προσελκύσει επενδύσεις οφείλει να έχει μία ενέργεια, μία μάλλον μετάβαση ενεργειακή που θα ορίζει σαφώς τα πράγματα. Γιατί αυτή η νομική βεβαιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Διακόπη. Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ πολύ. <laughs> Εντάξει, τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο να τελειώσετε το λόγο σας 1,5 λεπτό, αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα, εδώ τελειώνει ο κατάλογος ε, των εισηγητών και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρόιλ. Και εγώ κάποια πολύ σύντομα σχόλια έχω να κάνω. Καταρχάς, αν θέλουμε πρόοδο, όπως είπε ο Κλοντ, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει οικονομικά. Αλλά αυτό χρειάζεται και αποδοτικά μέτρα. Δηλαδή, χρειάζεται συνέπεια, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να είμαστε ρεαλιστές και να μην ε, προβάλλουμε ε, υπερβολικές απαιτήσεις. Ο κατάλληλος τρόπος ε, σίγουρα δεν είναι με γραφειοκρατία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ο καθένας τη δική του δυναμική, τις δικές του ιδιαιτερότητες. Και το καλύτερο θα ήταν εάν δώσουμε έμφαση στην αποδοτικότητα και αν ε, ακούσουμε τις απόψεις των διάφορων ομάδων ενδιαφερομένων. Και φυσικά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα πολύ καλό και λειτουργικό σύστημα ελέγχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πολύ με τα όσα ανέφερε ο κύριος ε, Τούρμες. Όταν μία επιχείρηση με τα χρήματα της ίδιας τράπεζας ε, σε δύο διαφορετικά κράτη-μέλη ε, δηλώνει τελείως διαφορετικές επενδύσεις, μάλλον πρόκειται για απάτη, γιατί ε, προσπαθεί να αποκτήσει και να εξασφαλίσει επενδύσεις ε, υψηλότερες, ε, όμως πρέπει να θεσπίσουμε όρια, δηλαδή αναγνωρίζουμε το υψηλό κόστος των επενδύσεων στο κατάλληλο όμως επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα επέτρεπε να συνδέονται απευθείας ε, το κόστος ε, στο πραγματικό κόστος κεφαλαίου και από την άλλη δεν δίνουμε έτσι κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις ε, να κάνουν τέτοιες μη ρεαλιστικές δηλώσεις κεφαλαίων. Τώρα, Πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι ε, το ζήτημα αυτό αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίους και ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα σε αφορά την ενεργειακή ένδυα, ότι αυτό ε, πλήττει 70 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Μετά, Πρέπει να εξετάσουμε όλο τον ε, κύκλο, όλο το πλαίσιο της ενεργειακής ε, αγοράς και τους παρόχους και τους παραγωγούς και τους διανομή. Ε, γιατί εκεί στη διανομή έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό απολειών Πρέπει λοιπόν να πούμε πού ακριβώς υπάρχουν αυτές οι απώλειες, πού αποκρύπτονται ορισμένες δαπάνες και πού τελικά ε, επομίζονται οι καταναλωτές, οι εμπορευόμενοι. Πρέπει εμείς να δώσουμε την απαραίτητη έμφαση. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Γκροστέτ. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι το κείμενο αυτό για την διακυβέρνηση είναι κεντρική σημασία ε, που θα μα επιτρέψει να κάνουμε μια διασύνδεση μεταξύ των μέρου ε, εγγράφων για την ενέργεια. Για τη διακυβέρνηση πρέπει πάντα όμω να λαμβάνουμε υπόψη και τη βούληση των κρατών μελών. Υπάρχει λοιπόν κάποια ευελιξία ούτω ώστε ε, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τα δυνατά τους σημεία να αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό αντιστοίχως. Υπάρχει και ένα θετικό σημείο στα εθνικά σχέδια που προτείνει η Κομισιόν. Αυτό είναι ε, οι διαδρομές ανάτεχνολογία που θα παρουσιάζουν τα κρατημέλη. Αυτό επιτρέπει στην κρατημέλη να επιλέξει τον κλάδο της βιομηχανία που θέλει να ευνοήσει βάσει των ιδιαιτεροτήτων της ε, χώρα αυτής. Αυτό φαίνεται καλό και ήδη χθε και στην ακρόαση που κάναμε χθε το απόγευμα το ανέφερα στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ε, πρόσκληση υποβολή ενδιαφέροντος για κάθε συγκεκριμένο κλάδο και όχι για τεχνολογίες, γιατί ε, αυτές οι προσκλήσεις μπορούν ακριβώς να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Αλλά πραγματικά επιμένω σε αυτό και θα μείνω εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το είπαν αρκετοί, αλλά θέλω και εγώ να τονίσω ότι το ενεργειακό πακέτο είναι πακέτο, είναι δέσμη μέτρων. Ε, μέτρων που ε, συνδυάζονται. Γι' αυτό η Επιτροπή μας, μαζί με άλλες επιτροπές, δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό. Η διακυβέρνηση είναι το τελικό κομμάτι του παζλ, το κομμάτι που μπορεί να συνδέσει όλα τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια. Έχω να πω τα εξή σχετικά με την διακυβέρνηση. Ε, πρώτα, οι σκιώδει ηγητέ το είπαν, αλλά θέλω κι εγώ να αναφερθώ στην ενεργειακή ένδυα ως ε, στόχο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα εθνικά ε, ενεργειακά σχέδια να συμπεριλαμβάνουν και μάλιστα σε περίοπτη θέση το θέμα της επίλυσης ενεργειακής ένδυας. Έπειτα, ε, όπως είπε και ο συγκητής, η συνδεσιμότητα, οι διασυνδέσεις, η χωρητικότητα είναι απίστευτα σημαντικά. Η διακυβέρνηση εδώ ε, συνδέεται άρρηκτα με αυτό. Μετά, νομίζω πως ε, δίνουμε πολύ έμφαση στα κράτη-μέλη και αυτό το κάνουμε με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η Ευρώπη, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, Βρυξέλλες και μετά τα κράτη-μέλη. Όμως, ο σημαντικός, ο σημαντικότερος ε, παίκτη είναι οι πολίτες, οι χρήστες, οι πολίτες μας και πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες, οι πολίτες θα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τα κράτη-μέλη, διότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεβαντόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπαν οι αγαπητοί Κάρινς και Χόκμαρκ, συνάδελφος. Συν... Σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα δείχνει μεγάλη δημιουργικότητα στην ε, δημιουργία και τροποποίηση κανονισμών, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από αυτό. Έχουμε το, την, το backloading, frontloading, έχουμε τις διάφορες αυτές ε, μεγάλες νομοθετικές πράξεις, αλλά ας ε, σκεφτούμε και σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα, πενταετή σχεδιασμό ας πούμε. Μετά υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία, υπερβολική γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στην Κομισιόν και μπορώ να φανταστώ τη δημιουργία μιας ε, ειδική υπηρεσία, η οποία να ε, ελέγχει ακριβώς αυτό, το ότι έρχεται από τα κρατημέλη, την γραφειοκρατία. Έπειτα, χρηματοδότηση. Μιλήσατε για μια πλατφόρμα χρηματοδότησης που ε, θα τροφοδοτείτε από τις επιδόσεις. Νομίζω πως ε, υπάρχει μία τάση να προσπαθούν τα κράτη-μέλη απλά να αποφύγουν την τιμωρία της ποινές που επιφέρουν οι χαμηλότερες επιδόσεις του επιθυμητού. Αυτό δεν είναι όμως στόχος δεν πρέπει να ε, υπάρχει αυτό το καρό των κονδυλίων που το οποίο προσπαθούν να φάνε τα κρατημέλη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κορουμπάτσεφ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω καταρχάς ότι, όπως είπε και ο Κλόντι, χρειάζεται απόδοση κεφαλαίου, όπως είπε και ο Κλόντ από ένα κιλοβάτ ε, στο Λουξεμβούργο μπορεί να παράγεις 900 κιλοβατόρε αλλά αλλού 400 κιλοβατόρε. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές λοιπόν, κάποιες ε, εγκαταστάσεις είναι αποδοτικότερε και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Χρειάζονται ανάλυση. Να πω τώρα ότι... ότι στη χώρα μου Βγήκε ο κόσμο στου δρόμους γιατί το κόστος της μεγαβατόρα ε, από ανανεώσιμες ήταν 360 ευρώ. Ο κόσμο βγήκε στους δρόμους, χαμό έγινε και η κυβέρνηση κατηγορήθηκε. Όλα λοιπόν τα κίνητρα για την πράσινη ενέργεια στη χώρα μας ε, είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Ο νόμος ε, εμποδίζει τα πάντα. Μίλαμε για φιλόδοξους στόχους, για 20, από το 27% στο 100%. Κάποιοι είναι πιο φιλόδοξοι, λένε ας μην μείνουμε στο 27, 30, 40, 50%. Και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα παζάρι στην Κωνσταντινούπολη και ψωνίζουμε χαλιά. Δεν υπάρχει και πολύ Κωνσταντινούπολη από την πατρίδα μου, 200 χιλιόμετρα μόνο. και τα ξέρω αυτά. Αλλά κάθε ποσοστό επί της 100 κοστίζει, κοστίζει χρήμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι φιλοδοξίες μας θα είναι και οικονομικά εφικτές. Ναι, και, και εμένα μου αρέσει να μένω σε ένα σπίτι 500 τετραγωνικών, αλλά, αλλά ε, η τσέπη μου αντέχει 100, τι θα κάνω. Μετά η Κάθλιν Φαν Πρέμπτ ε, είπε κάτι και θέλω να απαντήσω. Ναι, όταν η Γερμανία ας πούμε έχει ένα στόχο χ είναι στόχο τον οποίο νομίζει εκείνη πώ ε, θα επιτύχει. Δεν ισχύει αυτό για όλε τι χώρε. Α αφήσουμε λοιπόν τι ε, κοινέ ε, υποχρεώσει. Νομίζω πω αν υπάρχει μια κοινή υποχρέωση θα υπάρξουν προβλήματα. Γιατί μπορώ να σα πω από τη δική μα άποψη ότι ε, πολλές φορές σε ορισμένες περιφέρειες αν δεν υπάρχει ένας ε, υποχρεωτικό στόχο, περιμένουμε του άλλου πρώτα να κάνουν κάτι, λέμε πως εμεί δεν μπορούμε. Εγώ νομίζω πω και για την ενεργειακή απόδοση και για τις ανανεώσιμε χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι. Για όλους. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να έχει ζητήσει το λόγο. Α, ναι. Συγγνώμη, θα δώσω το λόγο σε εσάς. Ναι, ε, είχα ζητήσει το λόγο, συγγνώμη. Ε, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι που θεωρώ ε, ότι πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Εδώ δεν θέλουμε μόνο να είμαστε φιλόδοξοι, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Εφόσον όλοι χειροκροτήσαμε τα όσα επιτεύχθησαν στο Παρίσι, θα είμαστε υποκριτές εάν δεν εργαστούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ε, άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δύο, τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ε, ενέργεια και περιβάλλον. Ε, γιατί η επίτευξη αυτών των στόχων είναι θεμελιώδη. Ω εισηγητή τη έκθεση για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ε, ο προβληματισμό μου επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών και στο να είναι πιο φιλόδοξοι από αυτού που προτάθηκαν ε, ο στόχοι στο Παρίσι και για να είμαστε συνεχείς με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες με αποτελεσματικότητα και διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν κατά τη γνώμη μου η πρόταση διακυβέρνησης δεν προσφέρει σαφή συμβιβασμό που να εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί και με αδύναμη διακυβέρνηση και χωρίς δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο κάθε χώρα στην περίπτωση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της ε, μείωσης της χρήση του άνθρακα στο, ενεργειακό, στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον κύριο Τούρμες και για τροπολογίες θα υποβάλω και εγώ κάποιες και επίσης έχω την πρόθεση να ανακτήσω τους δεσμευτικούς στόχους ανά χώρα που είναι στην σημερινή οδηγία και που έχουν λειτουργήσει ε, αρκετά καλά και που δεν θέλω να ε, εξαλειφθούν από τις επόμενες οδηγίες. Ε, τα κατημέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε το γενικό στόχο, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό, κύριε Χούντ ε, Τούρμε, σε προτείνω να συντονιστούμε ώστε να ενισχύσουμε τόσο τη διακυβέρνηση όσο και την οδηγία για τις ανανεώσιμες ε, μαζί με την ε, ενεργειακή απόδοση και όπως είπα να πετύχουμε έτσι τους ε, στόχους. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος από ό,τι κατάλαβα αυτή τη φορά εξ ονόματος ε, εσάς του ιδίου. Ναι, μάλιστα. Μιλάμε για το κλίμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά δεν θα ήθελα διόλου να πω οτιδήποτε αντίθετα με την επίδευξη του στόχου. Απλώ θέλω να μιλήσω και για τους καταναλωτές που είναι σημαντικοί γιατί είναι και αυτή αντικείμενο της Ενεργειακής Ένωσης και όταν μιλάμε για καταναλωτές μιλάμε για κόστος και όταν σκεφτούμε πώς θα πρέπει να διακυβερνηθεί αυτό το σύστημα με τις εκθέσεις και ούτω καθεξής θα ε, διάβασα όσα είπε ο Γκούναρ και συμφωνώ μαζί του. Όταν σκεφτούμε το κόστος, ο Γκούναρ είχε μια σοφή πρόταση, αλλά νομίζω ότι ο βασικός νόμονας πρέπει να είναι ότι τίποτα δεν θα πρέπει να μπει περισσότερο εκτός αν και αν κάτι διαγραφεί. Είναι κάτι ε, που είναι πολύ εύκολο να θυμόμαστε και είναι μια κατευθυντήρια γραμμή ώστε να μειώνουμε το φόρτο. Γιατί τελικά ο καταναλωτής πληρώνει την ύφη. Και ο καταναλωτής είναι επίσης αυτός ο ίδιος που μας ψηφίζει. Uh, great time uh, Ναι, ναι, σπουδαίο αυτό που είπατε, γιατί ο έβδομος ε, εισηγητής για τη δέσμη της ενέργειας ε, είναι εδώ ε, στην αίθουσα, δεν έχει ακόμα καθίσει, αλλά είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Εφτά εισηγητές παρόντες στη συζήτησή μας, πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι περάσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι δική σας πρόταση. Νομοθετικές προτάσεις όλες περιχόνται από εσάς. Και ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεβόστ που είναι η Γενική Διευθύντρια της DG Ενέργεια. Γενική Διεύθυνση Ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζε, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τους εισηγητές και τους κοιόδες εισηγητές για τη δουλειά που έχουν ήδη κάνει. Θέλω να τονίσω κάποια σημεία τώρα και Καταρχά να πω προβλεψιμότητα και βεβαιότητα των επενδυτών. Είναι η εστίαση που δίνουμε στη διακυβέρνηση για την Ενέργεια και Ένωση, γιατί θέλουμε να υπάρχει περισσότερη προβλεψιμότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα σαφέ σημείο εκκίνηση για του ιδιώτε, αλλά και για, για το πακέτο ολόκληρο, με συγχωρείτε, αλλά και για την διακυβέρνηση. Επίση, καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια ώστε να ευθυγραμμίσουμε όλε τι υποχρεώσει αναφορών και δεδομένων ε, για όλες τις οδηγίες. Έχουμε εξετάσει όλες τις εκθέσεις, όλα τα σχέδια, τα προγράμματα των κρατών μελών και της Κομισιόν και τα εξετάσαμε ένα-ένα να δούμε ε, κατά ε, πόσο πρέπει να διαγραφούν γιατί έχουν ξεπεραστεί, πόσο πρέπει να ευθυγραμμιστούν και, και αυτό που προτείνουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα. Από τις 90 υποχρεώσεις περί ενέργειας, 20 τις καταργήσαμε, άλλες τις ολοκληρώσαμε, τις εντάξαμε ή τις ευθυγραμμίσαμε. Και πολύ λίγες τεχνικές θα μείνουν. Τεράστια προσπάθεια καταβάλαμε για να ευθυγραμμίσουμε την υπάρχουσα, τον υπάρχοντα σχεδιασμό και τις αναφορές ώστε να έχουμε λιγότερο διοικητικό φόρτο. Για παράδειγμα για τα εθνικά πλάνα αποδοτικότητας και τα εθνικά πλάνα για τις ανανεώσιμες από το 2020 θα περιλαμβάνονται στα ολοκληρωμένα εθνικά προγράμματα. Πολύ, πολύ ε, συντονισμός λοιπόν. Τώρα, για τα εθνικά πλάνα ο εστιασμός δίνεται στο 2030 για τους στόχους, για το αέριο του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες κτλ. Χρειάζεται η διακυβέρνηση να είναι φιλόδοξη, οι ευρωπαϊκοί στόχοι να ακολουθήσουν όσον αφορά το σχεδιασμό και τις αναφορές από την πλευρά της Κομισιόν. Αλλά καλύπτουμε και όλες τις επιτυχές της Ενεργειακής Ένωσης. Σημαίνει κάποιες από αυτές τις αναφέρατε μόλις υποδομές, ενεργειακή φτώχεια, βεβαίως πολύ σημαντικός τομέας. Ε, στο ίδιο το πακέτο έχουμε διάφορα στοιχεία όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση αλλά θα ακολουθήσει και στην πρόταση περί διακυβέρνησης. Και κάτι ακόμα που ανέφερε ο Κλοντ και άλλοι είναι η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Θέλουμε το εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις να συγκεντρώσουν και να εμπλέξουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς από τη βιομηχανία τους πολίτες, τους καταναλωτές, εθνικές κυβερνήσεις, ε, όλους, όλους. Αυτό το έχουμε ήδη βάλει στα αιτήματά μας και επίσης να διαβουλευτούν και με τις ε, γειτονικέ χώρες. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που θα δώσουμε συνέχεια. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τα κάθε μελη στην τεχνική προετοιμασία, γιατί πρέπει να γίνει και τεχνική δουλειά για όλα αυτά. Σίγουρα όμως είναι σημαντική πτυχή. Τέταρτη παρατήρηση, περιφερειακή συνεργασία αναφέρθηκε με τον Κλόντ. Ήδη έχουμε κάποια καλά παραδείγματα όπου έχουμε δείξει στο, στις μας εκτιμήσεις αντικτύπου Έχουμε δείξει τις οικονομίες κλίμακας ε, που έχουμε κάνει. Το κόστος χαμηλώνει όταν ε, υπάρχει τέτοιο συντονισμός με τα κρατημέλη. Μπορούμε αυτό να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Εργαζόμαστε για τα στοιχεία που θα δείξουν τα κέρδη από την περιφερειακή συνεργασία. Έχουμε κάνει ε, τέτοιες ε, προσπάθειες, έχουμε δείξει ε, και έχουμε πάει πάρα πάνω και πέρα από το σημείο κίνησης των υποδομών και θα το ε, αναζητήσουμε ακόμη περισσότερο από την αναλυτική άποψη. Τελευταία μου παρατήρηση από κόστος, ωφέλεια και χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό, θέλουμε να συνοδεύσουμε ολόκληρη τη δέσμη με δημοσιονομικά μέσα, ας πούμε για ΕΦΗ, e, χρηματοδότηση για ΕΦΗ, e, κτίρια, αλλά έχουμε και προγράμματα περιφερειακά, έχουμε το ΕΦΣΥ, όπου δίνεται έμφαση στην ενέργεια και το κλίμα και όπου έτσι έχουμε ε, ένα σχεδιασμό που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος. Και αφήνω το λόγο στον συνάδελφο. Καλημέρα, να προσθέσω μόνο το εξή. Χάντε το μικρόφωνο το μιλητή. Here we are. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στο σχεδιασμό και τη στρατηγική Νομίζω ότι από την πρόταση γίνεται μια σαφής ε, διάκριση στη στρατηγική που είναι μακροπρόθεσμη και στο σχεδιασμό που είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για την επόμενη δεκαετία. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Άκουσα το επιχείρημα και εδώ αλλά και εκτός κοινοβουλίου ότι κατά κάποιον τρόπο πρώτα ε, καταρτίζουμε το σχεδιασμό και μετά τη στρατηγική. Από την ισχύουσα νομοθεσία και από τον κανονισμό σήμερα ήδη υπάρχει διάταξη για τα κράτη-μέλη κατάρτισης στρατηγικών. 11 κράτη-μέλη έχουν μια τέτοια στρατηγική και όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή τις ε, καταρτίζουν, τις προετοιμάζουν και βρίσκονται σε προωθημένο στάδιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι το 2020 θα πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμη στρατηγική, Απλώς ε, αυτό συνδέεται με τα όσα πρέπει να ε, υλοποιηθούν βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων και πρέπει να είναι έτοιμα το 2020. Όμως το σχέδιο που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για την ενέργεια και το κλίμα, είναι η πρώτη φορά που θα είναι ολοκληρωμένο σχέδιο, θα βασίζεται στις στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεκινάμε λοιπόν από το μηδέν. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και τον εισηγητή για τον κανονισμό Acer. Θέλατε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόμου τη κυρία Καρολίνα Πούνσετ, είμαι εδώ που είναι ε, για αυτό το φάκελο. Δεν μπορούσα να εδώ σήμερα. Θα ήθελα όμω για την άλλη να πω τα εξή. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για πρώτη φορά ζητά από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τέτοια ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Θεωρούμε ότι το νέο σύστημα διακυβέρνηση θα διευκολύνει τη διαμόρφωση εθνικών ε, πολιτικών αλλά και τη διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, χαιρετίζουμε το γεγονό ότι υπάρχει δεσμευτική πρόβλεψη για την προετοιμασία αυτών ε, και αυτό θα διευκολύνει την συγκρισιμότητα. Από πλευρά επενδυτών, λοιπόν, σίγουρα θέλουμε να μιλήσουμε, ε, να πούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη και για την ε, δημιουργία απασχόληση και την ανάπτυξη και κατά τη γνώμη μα απαιτείται και μία ε, αναφορά στα συγκεκριμένα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα προς τα κράτη-μέλη. Αυτή η διαδικασία θα αποτελέσει σημαντικό θεμέλιο για την ε, επίτευξη των στόχων μας, οπότε και η θέσπιση σημείων αναφοράς και για τις ανανεώσιμες αλλά και για την ενεργειακή απόδοση για να μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδο που θα σημειώσουμε είναι κέρια σημασία. Και τέλος, η υποχρεωτική συμμετοχή των ενδιαφερμένων μερών για μας είναι θετικό στοιχείο και θέλουμε να το τονίσουμε. Στα εθνικά σχέδια πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταρτίζονται μόνο από τεχνοκράτες, αλλά και από τους δήμους και κοινότητες. Να είμαστε κοντά λοιπόν στους πολίτες. Αυτά από πλευρά μα ε, και βεβαίω θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και τη συνεργασία. Πρόεδρο, η πρώτη συζήτηση είναι αυτή στην Επιτροπή Ήτρε. Βεβαίω ξεκινούμε με την διακυβέρνηση. Πριν ε, τα καταληκτικά σχόλια και τη σύνοψη από τον εισηγητή, ίσως θα ήθελε κάποιος να προσθέσει κάτι ή να ρωτήσει, γιατί είναι η πρώτη συζήτηση και έχουμε 7 εισηγητέ μαζί μας. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που βλέπω. Ο εισηγητή κύριο Τούρμα. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρούμπατσεφ για αυτό που είπε για τα χαλιά στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιες φορές, όντω μπορεί κάποιο να έχει την εντύπωση ότι ο καθορισμός ε, στόχων είναι σαν ένα παζάρι χαλιών. Λυπάμαι, αλλά όλα αυτά έληξαν το Δεκέμβριο του 2015. Με το Παρίσι έχουμε πλέον μία διεθνή υποχρέωση, 1,5 βαθμός. Μέχρι το 2050 μάλιστα πρέπει να φτάσουμε στο μηδέν Με τη φύση δεν υπάρχει τίποτα να διαπραγματευτούμε. Εάν περάσουμε το σημείο καμπής, τα πράγματα θα ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Και σας προειδοποιώ, όλους εσάς που δεν σας αρέσουν οι μετανάστες. Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να συμβεί. Και με, τα, το λέω και σε όλους αυτούς που λένε ότι είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Βλέπω κάποιους από αυτούς μπροστά μου. Τι προτείνουμε λοιπόν. Προεπολογισμό για τον άνθρακα, που είναι ο μοναδικός τρόπος να έχουμε μια επιστημονική, ακαδημαϊκή συζήτηση για το πού θα μπουν οι στόχοι το 2030. Ήδη τους έχουμε καθυστερήσει ε, εδώ και δεκαετίες. Έχουμε ήδη αργήσει λοιπόν. Προπολογισμό για τον άνθρακα και από το 2050 επιστρέφει στο 2030 και βλέπουμε τι είναι ρεαλιστικό. Οι καταναλωτές είναι σημαντικοί, αλλά πάνω απ' όλα είναι πολίτες θα είμαστε 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε έναν πλανήτη. Εάν δεν κινηθούμε γρήγορα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και υπάρχουν και καλά νέα. Κάναμε λάθη στη Βουλγαρία, στην Ισπανία. Στην Ισπανία είχαμε 450 ευρώ ανά κιλοβατόρα. 360 στην ε, Ρουμανία. Αυτό δημιούργησε μια κακή εντύπωση. Είχαμε το διαγωνισμό στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα για 55. Στη Δανία για 55. Είναι λοιπόν, ήταν μάλλον ε, ακριβές οι ανανεώσιμε. τώρα είναι φτηνές. Αν καταφέρουμε όμως να τα συνδέσουμε στα δίκτυα. Και, όσοι και προς τους υπέρμαχους των υπόλοιπων ε, πηγών ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια τώρα είναι δυόμιση φορές πιο ακριβή. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Όχι. Έχω, θέλω ακόμα ένα λεπτό. Το μήνυμά μου προς την Επιτροπή. Χρειαζόμαστε δράση αυτή τη στιγμή και από την Επιτροπή. Ποιες είναι οι ε, προτάσεις για τον προπολογισμό μετά το 2020. Διακόπτει ο Πρόεδρος και πάλι. Και η ιδέα του κ. Μόντι για, για τους ίδιους πόρους πρέπει να συνδεθεί εδώ. Έχουμε κάποια προσκόμματα, η δίκαιη μετάβαση. Έχει πεθάνει ο άνθρακας, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ένα μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται. Ενεργειακή ένδυα. Λυπάμαι, αλλά η φτώχεια είναι φτώχεια. Χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ε, κατάργησης της λιτότητας και με αυτό το ενεργειακό πακέτο μπορούμε να δημιουργήσουμε και θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Το χρονοδιάγραμμα τώρα, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης 21-22 22 ιουνιου κατάθεση συγγνώμη, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Ιουνίου. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος λοιπόν. 4 Σεπτεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα και ψηφίζεται τον Οκτώβρη 11 και 12 Οκτωβρίου στην Ήτρε. Επόμενο τώρα σημείο και πάλι στην ίδια δέσμη ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση. Εισηγητής ο κύριος Ανταμ Κίρικ. Ίδια είναι η παρουσίαση. Δεύτερο σημαντικό θέμα στην ενεργειακή δέσμη. Ξέρουμε ότι η ενεργειακή απόδοση είναι και ο τρίτος πυλώνας της Ενεργειακής Ένωσης. Πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Συνάδελφε Γκέρεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. η Επιτροπή με την πρότασή της για την τροποποίηση του κανονισμού του 2012 είναι λανθασμένες όμως ε, οι διαπιστώσεις, γιατί όλα αυτά οφείλονται στην ασφαλή ενέργεια και όχι στην απόδοση. Πράγματι οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας. Όμως η εξοικονόμηση στην αγορά δεν προκύπτει πάντα από την αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Πρώτα λοιπόν έχουμε διάφορες μορφές πρωτογενούς ενέργειας, πρωτεσίλες, ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες. Η πρωτογενής ενέργεια λοιπόν θα πρέπει να θεωρείται ως ε, πρωτογενής ενέργεια που συσσωρεύεται και έτσι αθρηστικά ε, αυτό μας επιτρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ενέργεια. Δεν είναι μόνο ο άνθρακας ε, που είναι το βλαβερό, είναι και ε, όλη η προσπάθεια που απαιτείται για την εξόριξη του άνθρακα. Με τα πυρηνική ενέργεια είναι πολύ δαπανηρή. Η πρωτογενής ενέργεια μετατρέπεται στην τελική μορφή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής. Ποιος πρέπει να είναι λοιπόν ο σκοπός της οδηγίας. Εάν διαφέρει από αυτό που μας παρουσιάζει η Επιτροπή. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση ε, των πρωτογενών ορυκτών καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η Όλα αυτά μπορούν να υπολογιστούν μέσω ε, της ανάλυσης του κύκλου ζωής. Έτσι έχουμε την επιλογή μεταξύ πρωτογενούς και τελικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός αυτός γίνεται λανθασμένα, γιατί η μείωση της πρωτογενούς ενέργειας δεν σημαίνει ότι περιορίζουμε την χρήση των ορεικτών καυσίμων. Σκοπός λοιπόν θα πρέπει να είναι ο περιορισμός των αθεριστικών πρωτογενών ορυκτών καυσίμων. Η μετατροπή λοιπόν της ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υπολογίζεται ως πρωτογενής και η χρήση ορυκτών καυσίμων. Υπολογίζουμε λοιπόν την πρωτογενή κατανάλωση και την ενέργεια που απαιτείται ε, ως απόθεμα σε περίπτωση που δεν υπάρχει άνεμος ε, ή ηλιοφάνεια. Η Επιτροπή θέλει να αναφέρεται μόνο στο τελικό στάδιο της χρήσης ενέργειας που είναι ηλιανική. Όμως έτσι εξεφεύγουμε από την ενεργειακή απόδοση. Μιλούμε περισσότερο για την εξοικονόμηση ενέργειας από τους καταναλωτές. Αυτό αφορά μόνο δηλαδή την ε, ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής που προσδιορίζεται πολύ συγκεκριμένα. Οι ευρωπαϊκές χώρες ε, σε τη αφορά κατακεφαλήν κατανάλωση ενέργειας και το ΑΕΠ μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι μέχρι τις 3.000 ε, ε, κιλοβατόρες κατά άτομο, μετά 5 έως 6.000 κιλοβατόρες ανά άτομο χρόνο και σε κάποιες χώρες είναι πάνω από 7. Βέβαια, με την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας αυξάνεται και το ΑΕΠ. Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε την ενεργειακή απόδοση ως ε, περιορισμένη κατανάλωση μέχρι το 2020 μέχρι το 2030. Μπορεί να γίνει αυτό σε όλες τις χώρες. Κάποιοι λένε ότι θα είναι και ως 40% μέχρι το 2030, βέβαια σε σχέση με το έτος αναφοράς. Υπάρχει λοιπόν ένα ξεκάθαρο ζήτημα. Αυτή η νέα οδηγία ενεργειακής απόδοσης πώς θα πρέπει να συνδέεται με τη νέα οδηγία για το ETS. που καθορίζει τις τιμές κατανομής εκπομπών. Η οδηγία λοιπόν ETS θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση ό,τι αφορά την πρωτογενή ενέργεια, που είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τον ορισμό που δώσατε στην ενεργειακή απόδοση, ότι είναι δηλαδή η ενεργειακή απόδοση των πρωτογενών πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση. Πρώτος θα λάβει το λόγο εκ μέρους του ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε μόλις τώρα από τον ε, συνάδελφο Τόμας ε, είναι καταστροφικά. Μας λέει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι πρωταθλήτρια. Έχει χρυσό μετάλλιο σε οτιδήποτε αφορά το περιβάλλον. Ε, εξοικονόμηση ενέργειας, ε, ε, μείωση διοξιδίου του άνθρακα ανανεώσιμες. Είμαστε μάλιστα τόσο καλοί που η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση έχει τεθεί σε ισχύ α, πολύ καιρό και μάλιστα επιτύχαμε τους στόχους του μείον 20% το 2014. Υπάρχουν ορισμένες δεσμευτικές υποχρεώσεις που έχουμε εδώ και δεκαετίες και ε, νομίζω πως ε, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, δεν έχω κάποια γυάλινη μαγική σφαίρα, όμως σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή και με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις προσπάθειες για αυτούς τους στόχους. Τώρα, ε, εγώ είμαι υπέρ του 30% και μπορώ να επιχειρηματολογήσω υπέρ αυτού. Αυτός ο στόχος όμως χρειάζεται επανεξέταση και ενδεχομένως αναπροσαρμογή κάθε δύο-τρία χρόνια. Και εάν δεν υπάρχει δεσμευτική, δεσμευτικό σε 1,5% για κάθε κράτος μέλος, τότε θα τεμπελιάσουμε. Είμαι τώρα της άποψης ότι το άρθρο 7 πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, πρέπει να υπάρχουν ακόμα περισσότερα εναλλακτικά μέτρα και θεωρώ επίσης ότι οι δράσεις που έχουν προταθεί δεν νομίζω πως ανταποκρίνονται πλήρως ε, στις φιλοδοξίες μας. Από την άλλη βέβαια, είμαι λίγο χαλαρό, γιατί νομίζω πω δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι τόσο περίπλοκα, αρκεί να επικεντρωθούμε σε αυτά τα τρία άρθρα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και α μην κάνουμε του ξερόλε εδώ στο Κοινοβούλιο, α μην δημιουργούμε νέα άρθρα και ε, αναδεύουμε τα πάντα. Α επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό. Υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Ε, μάλιστα η αριστερή πλευρά του Κοινοβουλίου έχει προτείνει ένα στόχο του 40%. Αυτό πιστεύω πως ε, δεν είναι εφικτό. Είναι καταστροφικό. Ε, θα αλλάξουν τα πάντα. Θα έρθουν τα πάνω κάτω με την αγορά. Θα ανακληθούν άδειε επιστοποιητικά εκπομπών κτλ. Όμως ε, νομίζω πως κάθε περίπτωση με τους σκιώδεις και με τον εισηγητή θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Βαν Πόσουιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να πάρω το λόγο για αυτό το φάκελο, για την ενεργειακή απόδοση και που έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκάθαρα ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να έχει προτεραιότητα. Σε τη την Ενεργειακή Ένωση. Υπάρχουν όμως και κάποιες σκέψεις που έχω και προβληματισμοί σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα τον σκοπό της αποδόσης που είναι το 30% στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς όμως θα κατανοηθεί αυτό το 30% ε, στα κράτη-μέλη και πώς έτσι θα επηρεαστούν τα κράτη-μέλη κάνει λόγο για 400.000 θέσεις απασχόλησης η Κομισιόν, αλλά πού θα δημιουργηθούν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτήματα γύρω από αυτούς τους στόχους και στηρίζω ε, και το όραμα που έχει προωθήσει η δική μου περιφέρεια, η Φλάνδρα, ε, στο Συμβούλιο μεταξύ των κρατών μελών, όπου ζητούμε πρώτα απ' όλα περισσότερες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο ε, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ε, ε δεσμευτούμε για συγκεκριμένα ποσοστά. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, εγώ επιμένω στο 27% όπως έχει οριστεί στο Συμβούλιο το 2014. Επίσης, νομίζω ότι πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία μέτρα του παρελθόντος που έχουν ε, ε, μακροπρόθεσμο αντίκτυπο να μην λαμβάνονται υπόψη. Γιατί υπάρχει και ε, ζητούμε μάλλον 1,5% κάθε χρόνο προσθετικά, όμως ποιος θα πληρώσει το κόστος για όλα αυτά τα μέτρα, ποιος θα αναλάβει τις διαρθρωτικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αυτός είναι ο δεύτερος προβληματισμός και κάτι τελευταίο. Σίγουρα και η Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες ε, πληροφορίες. Ε, νομίζω ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία μάλλον θα πρέπει να υλοποιούνται όλο και περισσότερο από μια δυσανάλογη υποβολή εκθέσεων και διάφορα μαγικά, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ξεκάθαροι και σαφέστατοι κανόνε για τα κράτη-μέλη για την υποβολή εκθέσεων, τι ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και τι όχι. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό την πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή για τη διακυβέρνηση ε, να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και έτσι δεν έχει πολύ νόημα να εφαρμόζονται, να επιβάλλονται μάλλον δεσμεύσεις και υποχρεώσεις προς τα κράτη-μέλη ήδη να έχουν ένα πρώτο εθνικό σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια το 2018. Εδώ τώρα συζητάμε εμεί του στόχου. Πώ γίνεται το 2018 να υπάρχουν και έτοιμα εθνικά σχέδια. Όμω ε, έκανα μια πρώτη συζήτηση με τον εισηγητή, πολύ ε, ενδιαφέρουσα και θέλω να συνεχίσουμε αυτήν ακριβώ τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Θα σα ζητήσω την επόμενη φορά να είστε πιο σύντομο. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι βέβαια. Ε, κύριε Τούρμε, έχετε το λόγο. Εκ μέρου των Πρασίνων, φυσικά και όσο αντικατασ... το κύριο του κύριου Γιάβορ. Ναι, ο κύριο Γιάβορ δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να καταστραφεί η ασφάλεια και η σιγουριά των επενδυτών με το να υπάρχει αυτή η ρήτρα για το 2030. Τι έχουμε κάνει με την τελευταία οδηγία ε, περί ενεργειακής απόδοσης. Ήμουν και εισηγητής αυτή. Δημιουργήσαμε αγορές ενεργειακής απόδοσης. Το χειρότερο μπορεί να κάνετε σε έναν επενδυτή είναι να του πείτε ότι υπάρχει αγορά, η αγορά όμως αυτή τέρμα, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει. Και θεωρώ ότι η ανάλυση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν πρότεινε αυτή την άδεια πάυσης κυκλοφορίας, είναι να καταλάβει ότι για να διατηρήσουμε αυτή την αγορά ενεργειακής απόδοσης πρέπει να σταματήσουμε πλέον να χρησιμοποιούμε αυτή τη ρήτρα. Να σας τα πω και στα γερμανικά κιόλα, ε, κύριε συνάδελφε. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο για το περιβάλλον που έχει εφαρμόσει η καγκελάριό σα, η κυβέρνησή σας και ψηφίσατε όλοι. Αν το θέλουμε αυτό, τότε πρέπει ε, να, να χρησιμοποιήσουμε απίστευτα τεράστια ποσοστά ενέργειας μέχρι το 2030. Όλοι όσοι ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα, με, το, με την κλιματική αλλαγή και έχουν δει τις διάφορες προβλέψεις, λένε πως η ενέργεια είναι το σημαντικότερο. Και γνωρίζουμε όλοι ότι ακόμα και μετά το 2030 πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για ενεργειακή απόδοση. Ε, και τι έχει κάνει, ας πούμε, α, η κυβέρνηση άλλου κράτους ή της Γαλλίας. Έχει βάλει στόχο μέχρι το 2050. Έχει ξεπεράσει το 2030. Μα δεν γίνεται αλλιώ. Διότι διαφορετικά, τι είναι αυτά που λέτε, πρώτα η ενεργειακή απόδοση, πρώτα το περιβάλλον. Μα κοροϊδεύεται. Χωρί να υπάρχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δεν γίνεται τίποτα. Και αυτέ οι αγορέ τι οποίε χτίσαμε με πολύ κόπο, με πολύ υπομονή, ε, κινδυνεύουν να καταστραφούν ακριβώ από αυτή τη ρήτρα παύση ε, άδεια κυκλοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Περίτο Λουάγκα εκ μέρους της ΓΚΟΕ έχει το λόγο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμά δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρωτοθλητές αν ε, δεν ε, καταφέρουμε να αποφύγουμε την κατάρρευση του κλίματος και ο τελευταίος ο οποίος βοηθά στην κατάρρευση είναι ο Ντόναλτ Τραμπ. Εμεί θέλουμε να ανακάμψει η οικονομία μέσω του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και, απα... και, και, και να εξοικονομήσουμε ταυτόχρονα ενέργεια πράγμα το οποίο έχει και κοινωνικά ωφέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για 40% μέχρι το 2030 γιατί κάθε ποσοστό παραπάνω που κάνουμε μας οδηγεί πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου. Ε, εάν θέλουμε να έχουμε διαφορετικό ορισμό ευρύτερο για τα ωφέλη και δεν βασιστούμε τόσο στο κόστος. Ο στόχο του 40% αντί για 30% αντιπροσωπεύει μια μείωση των εισαγωγών ε, φυσικού αερίου κατά 29%, 4,4 εκατομμύρια θέσεις επιπλέον απασχόλησης και καλύτερη, ε, ε, μάλλον και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Θα πρέπει να θεωρήσουμε την ενεργειακή μετάβαση ως ευκαιρία για να αλλάξουμε πρότυπο και μοντέλο και να διατηρήσουμε τους στόχους μας μακροπρόθεσμα και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να επιμείνουμε στο δεσμευτικό χαρακτήρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό και ελπίζουμε πως αυτό θα συμπεριληφθεί στην οδηγία περί διακυβέρνησης που ε, ε, συζητήσαμε προηγουμένως. Άρθρο 7 δε που θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά σε αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ευελιξία και τις νομικές ελλείψεις ε, ή κενά και για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η, λειτουργία θα, αυτή η οδηγία θα λειτουργήσει θα πρέπει να εξαλείψουμε κάθε παραθυράκι που ενδεχομένως να υπάρξει. Αυτά τα παραθυράκια ή τα κενά μέσω του τομέα της μετάφρασης, ε, της, των μεταφορών με συγχωρείτε, είναι αυτά που τελικά μπορεί να οδηγήσουν στην μείωση του από το 1,4% στο 0,1%. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταμπουράνο, εξ του EFDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε, αρκετέ φορέ έχουμε συζητήσει πόσο πολύ η, εθνη, ενεργειακή απόδοση είναι ένα στόχο πολύ βασικό. Είναι θέμα γεωπολιτικό για την ανεξαρτησία τη Ένωση από τα ρηκτά καύσιμα, βελτίωση οικονομική, ε, απασχόληση, κοινωνικές βελτιώσεις και καταπολέμηση των εγκληματικών αλλαγών. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Όμως θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται για μια δημόσια πολιτική που δημιουργεί ευκαιρίες. Πρέπει, μπορούμε να χάσουμε το τρένο ε, χωρίς να βάλουμε το πύχη πολύ ψηλά. Ε, γι' αυτό θέλ, θέλω να επαναλάβω την ανάγκη να φτάσουμε πάνω από το 40% που ορίζεται στους εμμονωμένους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Επίσης είναι τρελό να δίνουμε την δυνατότητα στα κρατημέλη από τη μια πλευρά να αποκλείουν την ολοκληρωμένη ενέργεια στον τομέα της, ε, των μεταφορών από τον υπολογισμό της τελικής ενέργειας που τελικά θέλουμε να φτάσουμε στο 1,5% και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά τα ίδια κράτη να έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τις εξοικονομήσεις που έχουν επιτύχει ε, μέσω των αλλαγών πάντα στον τομέα των μεταφορών που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Νομίζω πως αυτή η προσέγγιση δεν είναι και πολύ λογική και να τονίσω επιπλέον ότι από το 7-2 γράμμα ε απορρέει η δυνατότητα να αποκλειστεί από τον υπολογισμό ενεργειακής εξοικονόμησης η ενέργεια που παράγεται σε ε, τα κτίρια μέσα από τις πολιτικές που προωθούν την αυτοκατανάλωση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι ε, αυτός ο στρεβλός ο κανονισμός. Αντί να έχουμε δηλαδή το Energy Efficiency First, ε, δίνεται κίνητρο για την παραγωγή ανανεώσιμων ε, ενεργειών, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται παρκώς, με πάνελ που παράγουν δηλαδή ενέργεια που απλά σπαταλάται. Μήπως κάποιοι να εδώ τη δυνατότητα να καταγράψουν όλα αυτά και να σκεφτείτε ότι σε κάποιες χώρες όπως η δική μου, ορισμένα μέτρα πρόθεσης των ανανεώσιμων μπορούν και να θεωρηθούν ως μέτρα ενεργειακής επάρκειας ή αποτελεσματικότητας. Τέλος, στο 10 ε, α, νομίζω ότι θα πρέπει καλύτερα να ορίσουμε τα μέτρα για την πρόσβαση και τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων των στοιχείων των ε, ε, χρηστών. εάν κανείς σκεφτεί τη μεγάλη οικονομική αξία που έχουν. Σαφχάουζερ και μετά Τιόκα, εξ, του των συντηρητικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πείτε ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά ε, θα ήθελα να δείξω τα μέσα μιας βολονταριστικής πολιτικής. Εάν υποθέσουμε πως μια χώρα είναι θέλει να κάνει 23% ε, στο, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού το οποίο με τη σειρά του, ο, ο οποίος μάλλον με τη σειρά του δυστυχεί στο 4% του ΑΕΠ. Δηλαδή να εξοικονομήσει το 1% του ΑΕΠ. Για να εξοικονομήσει κανείς το 1% του ΑΕΠ, το εγχώριο προόντο, σημαίνει 10% επενδύσεις και 10% ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωζώνης, που είναι γύρω 10, στα 13, θα έπρεπε να επενδύσουμε για να επιτύχουμε 103. Δηλαδή ένα, ένα τρεις επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν. Ναι. Λέμε στόχο, κάτι το οποίο απορρέει από μια φυσιολογική πολιτική, γιατί εδώ δεν υπάρχουν πραγματικοί νέοι στόχοι χωρίς νέα μέσα. Και αυτή η φιλοδοξία είναι προσβάσιμη, είναι προσιτή. Έχουμε την Κεντρική Τράπεζα που η οποία για κάποια χρόνια αγόραζε 1,5-3 ε, δημόσιο χρέος. Γιατί να τα αγοράζει το χρέος και να μην επενδύσει σε πραγματικές ε, υποδομές, γιατί αυτό θα με, μεταμόρφωνα την οικονομία, θα αντιστοιχούσαν ε, περίπου σε 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης επιπλέον και θα δίναν και μια, θα συμφιλίωναν την Ευρώπη με τις φιλοδοξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Έχουμε ακόμα δύο εισηγητέ εδώ στο κατάλογο, τον κύριο Μπλάνκο Λόπε, που είναι υπεύθυνο για την ανανεώσιμη ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο και πάλι. Η πιο φθηνή, πιο καθαρή και πιο ασφαλής ενέργεια είναι αυτή που δεν χρησιμοποιείται. Αυτό εξηγεί η πρόταση την οποία υποβάλλει η Κομισιόν θα πρέπει να εστιάσουμε στη βελτίωση της ε, ε, ε, έντασης της ενέργειας, γιατί αυτό μας φέρνει ωφέλη στην ασφάλεια, στην ενεργειακή ανεξαρτησία και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, αλλά και μειώνει τις εκπομπές. Μεγάλο κομμάτι αυτών των οικονομιών ε, μπορούν δε να καταπολεμήσουν και την ενεργειακή φτώχεια. Ωστόσο, υπάρχουν φράγμοι που εμποδίζουν κατά την άποψή μου την ανάπτυξη όλων αυτών. Ε, χρειάζονται πολιτικές για την πρόθεση όλων αυτών. Το, το είπαν και άλλοι ε, ομιλητέ ότι ο στόχο 30% δεν είναι αρκετά ρεαλιστικό και φιλόδοξο. Και επίση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κοινοβούλιο μα είχε, είχε ζητήσει 40% δεσμευτικό στόχο στο πλαίσιο τη ε, Συμφωνία του Παρισιού. Μεγαλύτερη φιλοδοξία και στόχοι για την ενεργειακή απόδοση θα επέτρεπε να έχουμε καλύτερη ποσόστοση όσον αφορά τον ενεργειακό ανεφοδιασμό από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όπως είπα, σε σχέση λοιπόν με την πρόταση διακυβέρνησης, σας προτείνω επίσης εδώ το, στο συνάδελφο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε την κατάργηση της χρήσης του άνθρακα με πιο αποφασιστικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα άλλο ένας εισηγητής είναι στον κατάλογο, ο κύριος Ζανονάτο, που είναι αρμόδιος για την προετοιμασία απέναντι στον κίνδυνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφέ σε όλους, το θύμισε μόλις και ο εισηγητής που μίλησε πριν από μένα ότι η απόδοση και η, οικονομική, ενεργειακή εξοικονόμηση είναι, είναι απαραίτητη ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού αλλά και για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή μετάβαση. Αυτά όλα θα πρέπει λοιπόν να είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας και πιστεύω πως ο στόχος του 30% είναι εξαιρετικά χαμηλός. Θεωρώ πως ο στόχος θα έπρεπε να είναι το 40%. Εκτιμάται ότι γύρω στα 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη θεωρούνται ενεργειακώς ευάλωτοι. Και αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τι ανατολικέ και μεσογειακές περιοχέ, τις νότιε περιοχέ τη Ευρώπη θα μπορούσαν και να αυξηθούν. Και γι' αυτό βρίσκω πω η αναθεώρηση του άρθρου 7 πρέπει να απαιτεί αυτή τη δέσμευση που είναι σημαντική για τα κράτη-μέλη, ώστε να περικόψουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή του κατανάλωση. Με την πρόταση τη Κομισιόν υπάρχουν ε, τι πτυχέ που δεν με πείθουν, Όμω, αυτό είναι το θέμα, το ένα είναι το θέμα τη ενεργειακή φτώχεια που θα πρέπει να οριστεί καλύτερα. Πρέπει να οριστούν οι δράσει οι ενέργειε που θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο στα θέματα ενέργεια. και ω προ αυτό, για παράδειγμα, υπάρχουν εμπόδια στα επενδύσει για την ενεργειακή απόδοση που θα πρέπει να αρθούν και ε, επίσης ε, θα πρέπει να αυξηθούν οπωσδήποτε τα κονδύλια που απευθύνονται στην ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μίκα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα επαναλάβω αυτά που είπα και προηγουμένως. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι απώλειες από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή είναι 15 έως 30% ανάλογα με τη χώρα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή την απώλεια την επομίζει το καθένα στο λογαριασμό του. Μπορεί κάποιο να πει ότι είναι απόλυτη προκύπτουν τεχνολογία, πώ να το περιορίσουμε. Αλλά αν ήταν έτσι, θα είχαμε τι ίδιε απώλειε σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω στην πράξη βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλε οι διαφορέ. Αυτό σημαίνει ότι ε, μια μείωση αυτών των απολειών από τον παραγωγό στον διανομέα, στον μεταφορέα μάλλον, στον διανομέα, ε, ανάλογα με τους ε, τρόπους αποθήκευσης ε, και τελική διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, τελικά θα μας οδηγούσε σε πολύ σημαντική εξοικονόμηση που θα μας βοηθούσε να πετύχουμε και το στόχο μας, δηλαδή να καταναλώνουμε λιγότερες πρώτες Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Στη Ρουμανία, οι μεταποιητές που έχουμε είναι πάρα πολύ παλιοί τι είδου ε, αποτελεσματικότητα και απόδοση να έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, όντω υπάρχει και κακή υλοποίηση, κακή συντήρηση έργων. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν δίκτυα τα οποία δεν είναι υψηλή τάση, αλλά μεσαία, το οποίο δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Σα δίνω λοιπόν παράδειγμα που θα μα ε, βοηθούσε να πετύχουμε τον τελικό μα στόχο. Στην άλλη οδηγία για την ενεργειακή αγορά θα πρέπει ο καθένας να έχει δυνατότητα να ε, βάλει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του και να παράξει έτσι ενέργεια. Γιατί αυτό θα είναι η καλύτερη μορφή ενεργειακή ε, απόδοση 100%. Ο καταναλωτής ε, θα καταναλώνει την ενέργεια που παράγει και όλοι θα είμαστε χαρούμενοι. Δεν περιμένω βέβαια απάντηση από την Επιτροπή ως προς αυτό το ζήτημα και ούτε άκουσα απάντηση γιατί τα φωτοβολταϊκά έχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με το χώρο, το μέρος δηλαδή, το οποίο δεν ε, δικαιολογείται από τις επιτυχίες τα λοιπά. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ παρότι που δεν απαντήσατε. Ευχαριστώ και εδώ στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς ε, όλου σα, λέει ο Μαχτά. Αυτό που δεν έχει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και η Ευρώπη είναι η συνοχή. Γιατί μιλούμε για ενεργειακή απόδοση, υπενθυμίζω σε όσους ε, έχουν αιμονή με το κόστος, ε, ο ενεργειακός λογαριασμό είναι 400 δις ευρώ το χρόνο. Ε, είναι πολύ σημαντικό κόστος λοιπόν για τις, και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Υπάρχει έλλειψη επενδύσεων μάλιστα το, τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει συνοχή λοιπόν. Χαίρομαι γιατί κάποιοι θυμούνται την COP21 στο Παρίσι, αλλά εδώ στρέφουμε προς την Επιτροπή, γιατί Ε, είχε κάνει και αυτές τις προτάσεις για το ETS. Υπερθυμίζω λοιπόν ότι η οδός που ακολουθήσαμε δεν ε, μας οδηγεί σε περισσότερες επενδύσεις, το αντίθετο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει ότι για να πετύχουμε τους ε, στόχους πρέπει να βάλουμε τον, την τιμή του άνθρακα των εκπομπών στα 190 δολάρια τόνο, που είμαστε πολύ μακριά από εκεί και θέλουμε, ε, ε, έχουμε το στόχο του 2,5% μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια συνοχή τουλάχιστον σε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ κυρία Γκρίφεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπε ένας συνάδελφος προηγουμένως ότι είμαστε ηγέτητα δύναμη στην καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ηγετική θέση. Η ενεργειακή ένδυα το παρατηρητήριο μάλλον γενετικής ένδυας ε, αυτή τη στιγμή δημιουργείται και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως πρέπει να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ όλων αυτών των τομέων και να τα εξετάσουμε όλα μαζί ως δέσμοι. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενεργειακή ε, απόδοση, είναι το πρώτο και κύριο. Και βλέπουμε ότι οι πιο φτωχοί ε, συμπολίτε μας είναι αυτοί που ζουν ε, στις χειρότερες συνθήκες. 50 εκατομμύρια λοιπόν σε ενεργειακή ένδυα. Από πλευράς επενδύσεων κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μακροπρόθεσμη βεβαιότητα για να έχουμε τις επενδύσεις που θέλουμε. Χρειαζόμαστε και δεσμευτικούς στόχους του 40%. Για παράδειγμα, με το στόχο του 27% γίνεται απόδοση 285 δις ευρώ στα ορυκτά καύσιμα, με το 40% 549. Τρία εκατομμύρια περισσότερα σπίτια μπορούν να ανακαινιστούν και 7 εκατομμύρια να ξεφύγουν από την ενεργειακή ένδυα. Πρέπει να βοηθήσουμε με υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξία του ενεργειακά φτωχού. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Να προσθέσω κι εγώ κάτι έτσι πολύ σύντομα. Ε, νομίζω δεν το έχουμε ακούσει πριν. Εάν ε, θέτουμε ένα και υψηλότερο στόχο ενεργειακή απόδοση, καταρχά πρέπει να δούμε αν τα καταφέρνουν τα κράτη-μέλη, αν μπορούν να τους ε, φτάσουν αυτούς τους στόχους. Ορισμένα κράτη δεν έχουν καν καταφέρει να εφαρμόσουν τους στόχους ε, που έχουν τεθεί μέχρι τώρα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ένδυα. Έχουμε ενδείξει ότι με τα μέτρα της ενεργειακής απόδοσης έγινε η κατασκευή κατοικιών ακριβότερη. Κοστίζουν πιο πολύ τα σπίτια τώρα. Και ε, όταν κοστίζει πιο πολύ να χτίσει ένα σπίτι, ανεβαίνουν και τα νίκια, οι άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλο εισόδημα δεν μπορούν να τα πληρώσουν και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μέτρο, τη μέση λύση, διότι ε, διαφορετικά οι, τα μέτρα αυτά θα έχουν ακριβώς τις αντίθετες επιπτώσεις. Οι πλούσιοι σίγουρα μπορούν να μένουν σε σπιτάρες, μονομένες κτλ. Οι άλλοι τι θα κάνουν όμως, πού θα μείνουν. Ας μην μιλάμε μόνο ε, θεωρητικά και μένουμε στα λόγια, ας δούμε στην πράξη τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you. I think in... Σας ευχαριστώ πολύ, κύριο Σκέλη. Νομίζω πως η ενεργειακή απόδοση είναι το ευκολότερο. Ο ευκολότερος στόχος που μπορούμε να πετύχουμε. Αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερες ενέργειες για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και να τους ενημερώσουμε για το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε δηλαδή ε, να μάθουμε στους πολίτες να ζουν ε, την καθημερινότητά τους με ενεργειακή απόδοση, ας πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν ενημέρωση. Και επίσης, όταν οι πολίτες πάνε να αγοράσουν μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένοι, να ξέρουν ποια από είναι η πιο ενεργειακά ε, όχι να πηγαίνουν και να επιλέγουν τη μάρκα που γνωρίζουν πιο πολύ από όλες τις άλλες, η οποία όμως ε, καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Εδώ βέβαια ε, πρέπει να συμπεριληφθεί και η συνεχόμενη διαβίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει όλοι να μαθαίνουν, να καταρτίζονται, να είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις και στον κατασκευαστικό τομέα και στην... στις οικοδομικές ε, υπηρεσίες, έτσι ώστε όταν κάποιος θέλει να, πάει, να αγοράσει ένα σπίτι, να μπορεί να επιλέξει την εταιρεία που θα το κατασκευάσει ε, και θα το κάνει πιο ενεργειακά αποδοτικό. Γι' αυτό λοιπόν η επαγγελματική κατάρτιση, η μάθηση είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κορουμπάτσοφ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να πω καταρχάς πως Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του κυρίου Γκίρεκ, να μην επικεντρωθούμε δηλαδή μόνο στην κατανάλωση, αλλά στην παραγωγή, τη μετάδοση και τη διανομή της ενέργειας. Οι απώλειες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά τα τρία επίπεδα είναι πολύ ψηλότερες από ότι ε, στο στάδιο της κατανάλωσης. Σίγουρα δεν πρέπει να χάσουμε ε, ε, το στόχο αυτό και να αγνοούμε την κατανάλωση, αλλά μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Δεύτερον, να σας φέρω και ένα παράδειγμα ενεργειακής απόδοση και σωστή προσέγγιση. Όταν παράγεις ε, θέρμανση από την ηλεκτρική ενέργεια. Στην δεκαετία του 90 όταν καταστράφηκε ένα εργοστάσιο που είχαμε παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναρωτηθήκαμε αν έπρεπε να το κρατήσουμε ή να το γκρεμίσουμε. Και ε, τι αποφασίσαμε, ότι καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια που θα κατα... να, το... να το καταστρέψουμε, αλλά την ενέργεια που θα χρειαστούμε γι' αυτό και την ενέργεια που θα παραχθεί να την ξαναδώσουμε πίσω ε, στο δίκτυο. Ή έτσι Είχαμε σχεδιάσει την ενεργειακή απόδοση και αυτή την εντύπωση είχαμε πως θα τα καταφέρουμε πριν από 20 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ενεργειακή απόδοση είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, ε, μεταφορών. Αν σκεφτούμε πόσα καύσιμα καταναλώνουν οι μεταφορές οι τα περισσότερα από αυτά είναι από ορυκτά καύσιμα. Επίσης, ε, πολλές φορές ε, χρησιμοποιούμε πυρημνική ενέργεια. Το κυριότερο πρόβλημα με τις μεταφορές είναι η κίνηση, ιδιαίτερα η κίνηση στα αστικά κέντρα και όταν πολλές φορές ε, βρίσκεις ουρές από γιοταχή ή φορτηγά οι οποίε ε, με, πάνε από φανάρι σε φανάρι, τότε ε, τι θα κάνεις, θα πηγαίνεις με πρώτη Δευτέρα, φρένο γκάζι, έτσι καταναλώνει περισσότερη βενζίνη, ανεβαίνει το κόστος της ε, ενέργειας. Υπάρχουν κάποιες καινοτόμες τεχνολογίες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, με οπτικές σε να γίνεται η σήμανση στα φανάρια έτσι ώστε να υπάρχει ομαλή κίνηση των αυτοκινήτων, να μην κόλλανε στην κίνηση. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι και με το, και με το μέρος μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, καθώς και οι τοποθετήσεις του κυρίου Γκίρεκ. Καταρχάς, ε, προτείνουμε στην αναθεώρηση ένα θεσμευτικό στόχο 30% για το 2030. Είναι μια αποχώρηση από το 27% που είχε αποφάσισε το 2014 από το Συμβούλιο. Ο κύριος Εγκύρεκ ε, σωστά τα είπε και από την πλευρά της, ε, του εφοδιασμού είναι πολύ ε, σημαντικό, αλλά και από την πλευρά της ζήτησης. Προσφορά και ζήτηση λοιπόν. Υπάρχει άμεσο συσχετισμός, όπως επίσης υπάρχει άμεση σχέση της προσφοράς και της ζήτησης με το ΑΕΠ. Το ίδιο και για τις ανανεώσιμες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ σημαντικές. Υπάρχει λοιπόν ε, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ο, την ενεργειακή απόδοση Σωστά. Τώρα, ο στόχος του 30% τονίζουμε ότι είναι η πιο οικονομικά αποδοτική λύση. Θα δημιουργήσει περίπου 400.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Σε ποιους τομείς? Κυρίως ε, στον τομέα των οικοδομικών εργασιών, κατασκευαστικών, αλλά και στη βιομηχανία. Σα στείλαμε ήδη κάποια στατιστικά στοιχεία, κάποια νούμερα με τα χαρά να το ξανακάνουμε ακριβώς για το πώς ε, θα γίνει αυτός ο καταμερισμός ε, των θέσεων απασχόληση στα κρατημέλη. Επίσης γνωρίζουμε ότι ένα στόχος 30% θα μειώσει κατά 12% τις εισαγωγές φυσικού αερίου και θα εξοικονομήσει εκατομμύρια από την ε, εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και αυτά τα δισεκατομμύρια αν ε, πάνε πίσω πάλι στην οικονομία θα οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΠ κατά 0,2%. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, νομίζω πως ε, προσπαθούμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, απομακρύνοντας αυτή τη ρήτρα παύσης ε, ισχύω. Αυτή θα λήξει το 2020 και στη συνέχεια επιθυμούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις στο άρθρο 7. Όπως είπε όμως και ο κύριος Πίπερ, θα υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης. Στην πρότασή μας προβλέπεται για το 2028. Έγινε και μια συγκεκριμένη ερώτηση για το άρθρο 7 παράγραφος 2. Δεν αποδυναμώνει την ε, ενεργειακή απόδοση, αντίθετα μάλιστα θα ενισχύσει την ε, χρήση των ανανεώσιμων. Θα τονίσω επίσης πως υπάρχουν πολλές συνέργειες ανάμεσα στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές εδώ άλλωστε. Γι' αυτό μπορούμε να συνδέσουμε τις ε, αντίστοιχες οδηγίες. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ενεργειακή ένδυα. Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να ωφελήσει και να επηρεάσει θετικά την ενεργειακή ένδυα. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΕΦΣΥ. Μας ε, παρουσιάστηκε και το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά. Τώρα, για το άλλο που είπατε, με την ενεργειακή αποδόση, εδώ υπάρχει και οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα κράτη-μέλη ε, έχουν τους δικούς τους ορισμούς για το τι είναι ενεργειακή ένδυα και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης έχουμε αποφασίσει να συσταθεί ένα παρατηρητήριο το οποίο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ενεργειακή ένδυα και θα κάνει σχετικές αναλύσεις. Και το, η ενεργειακή δέσμη μέτρων συμπεριλαμβάνει υπολογισμού για το κόστος της ενέργειας. Εδώ βλέπουμε ότι τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχουν αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Μας επιβεβαιώνει λοιπόν αυτό ότι τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα πληρώνουν περισσότερα για ενέργεια. Τέλος, να απαντήσω στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Νίκα. Ε, θα επανέλθουμε στο μέλλον και θα σας απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και να είστε σίγουροι πως θα συνεχίσουμε την ε, καλή επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, υπάρχουν οι σχετικοί κανονισμοί. Ο κύριος Μπέντσεν είναι εισηγητής στην Επιτροπή μας για αυτό το θέμα στα πλαίσια του ενεργειακού πακέτου και θα τον καλέσουμε την επόμενη φορά στην Επιτροπή να μας παρουσιάσει την δική του έκθεση. Αλλά τώρα είμαστε ακόμα στην ε, ενεργειακή απόδοση και θα δώσω τώρα το λόγο για τα τελευταία σχόλια στον εισηγητή κύριο Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την εντύπωση ότι σε πολλά ζητήματα δεν ε, καταλαβαίνόμαστε. Μια παράδειγμα, από την αρχή είπα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ενεργική απόδοση εκεί όπου οι απώλειες είναι μεγαλύτερες. Ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, παραγωγή και την μεταφορά της ενέργειας. Εκεί είναι ε, που πρέπει να αναζητήσουμε την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Αν δείτε κατά μέσο όρο την μετατροπή πρωτογενούς ε, ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, εκεί η απόδοση φτάνει κατά μέσο όρο το 40%. 60% λοιπόν της ενέργειας χάνεται. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση ε, στα νοικοκυριά. Εκεί έχουμε ε, μικρότερες ε, απώλειες, η απόδοση φτάνει το 60-65%. Όμως και πάλι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι αρκεί αυτός ο στόχος. Έχουμε εδώ λοιπόν τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε την οδηγία του 2012, ούτως ώστε όλες ε, οι χώρες να έχουν ένα κοινό όραμα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δεν απορρίπτει την αύξηση ενίσχυση της ε, εξοικονόμησης και στο 40% ή και παραπάνω. Αν βρούμε τις τεχνολογίες για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας, για παράδειγμα, ε, στα αργοστάσια παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η στην πυρηνική ενέργεια η απόδοση είναι 30-35%. Ενώ στον άνθρακα είναι ήδη 45%. Στην αιωλική είναι 40 50%. Την καλύτερη απόδοση την βρίσκουμε στα υδροελεκτρικά, έως και 90%. Πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε αυτά υπόψη, γιατί εκεί έχουμε τις απώλειες, εκεί χάνουμε πόρους και έτσι πλήττουμε το περιβάλλον. Καλό λοιπόν και τους κοιόδης εισηγητές να διευρύνουμε εδώ το περιθώριο Ακόμα και να αλλάξουμε τον ορισμό ενδεχομένω της οδηγίας του 2012. Είναι λανθασμένοι αυτοί οι ορισμοί από επιστημονικής άποψης. Να φτάσουμε ακόμα και εκεί. Εγώ έτσι έχω ορματιστεί ε, τις εργασίες μας ως προς αυτήν την οδηγία. Βέβαια, η βελτίωση της απόδοσης απαιτεί πολλές επενδύσεις. Και εδώ συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν για το οικονομικό σκέλος. Πράγματι, ε, αυτά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Όμως, πρέπει να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν ε, αυτά τα μέσα. Ευχαριστώ. Είναι καλό που κάνετε αυτή τη ε, διάκριση στην εξοικονόμηση στην τελική κατανάλωση. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τα κτίρια. Υπάρχει μάλιστα και ξεχωριστή οδηγία γι' αυτό. που αφορά άλλα ζητήματα τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Τονίσατε ότι κατά τη μεταφορά ενέργειας ή και κατά την εξόριξη ε, πρώτων υλών σπαταλούμε πολλούς ενεργειακούς πόρους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αποτελέσουν τμήμα της δέσμης για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα κτίρια είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σημαντική λοιπόν η προσέγγισή σας. Ε, η κυρία Γενική Διευθύντρια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να δώσει κάποιε απαντήσει, όμω και εγώ θεωρώ ότι ε, χρειαζόμαστε περισσότερε συζητήσει για να δούμε πόσο μπορούμε να αλλάξουμε την τεχνολογία, τι, πώς μπορούμε να παραμείνουμε στην ε, βιομηχανία, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ε, αγοράς τελικά, αλλά και της προόδου της τεχνολογικής εξέλιξης. Και αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της Συνεργικής Ένωσης. Η τεχνολογία και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις από τις ε, επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας. Δεν ξέρω πώς όλα αυτά μπορούν ε, να ενταχθούν σε ένα ενεργειακό πακέτο, αλλά ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία και λέμε ότι η ενεργειακή απόδοση δεν αφορά μόνο την κατανάλωση, αλλά όλα τα στάδια της ε, αλυσίδας. Θα έχουμε και άλλη μία συνάντηση για την ενέργεια και με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα καλέσω όλους τους ε, εισηγητές. Θα κλείσουμε τώρα την ε, συζήτηση για την ενεργειακή απόδοση του κυρίου Γκίρικ. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στις 21 και 22 Ιουνίου Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 28 Ιουνίου. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 4 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχες προθεσμίες όπως και για τη διακυβέρνηση. Ωραία. Τώρα ας περάσουμε στο σημείο 17. Όπως ξέρετε έχουμε καθυστερήσει 20 λεπτά. Αλλά ήταν φυσικό. Uh, συνάδελφοι, το επόμενο σημείο. Προαγωγή τη σύνδεση στο διαδίκτυο στι τοπικέ κοινότητε. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Συνδεσιμότητα στις τοπικές ε, κοινότητες. Ο συνάδελφος Κάρλος Ορίνιο είναι ε, εισηγητής. Παρακαλώ συνάδελφοι, Οι ιδιωτικέ συζητήσει να γίνουν εκτός της αίθουσας, παρακαλώ. Βέβαια, προτιμούμε να μείνετε μαζί μα, αλλά εάν δεν μπορείτε να μείνετε μαζί μα, παρακαλώ. Αποχωρήστε ησύχω. Ωραία, ξεκινήσουμε. Συνάδελφε Ζωρίνιο πολύ σημαντική έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Συνδεσιμότητα στις τοπικές κοινότητες. Ο κ. Ζωρίνιο στις 17 Φεβρουαρίου παρουσίασε το προσχέδιο έκθεσής του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Look like draft report. Τα έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η ημερομηνία, η προθεσμία μάλλον για την υποβολή τροπολογιών ήταν η Δευτέρα Μαρτίου. Τρέχοντος, δηλαδή. Και μέχρι τότε έλαβα 108 προτάσεις τροπολογίες μπορέσαμε έτσι να καταρτήσουμε 13 συμβιβαστικέ τροπολογίες που αφορούν την γενική φιλοσοφία της πρωτοβουλία αυτής, Τρει συμβιβαστικέ για την ε, εφαρμογή. Έγινε ήδη μία πρώτη σύσκεψη των ε, σκιωδών, ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι υπήρχε μεγάλη συνοχή σε σχέση με αυτήν την συμβιβαστική. Κατά βάση, με αυτές τις ε, συμβιβαστικές επιλύσαμε κάποια ζητήματα που ήθελα να υπογραμμίσω. Υποκαταστήσαμε μάλλον την έννοια της ε, δοτερότητας του δικτύου με την πιο κατάλληλη έκφραση του Open Internet Access, δηλαδή ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ. Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι το Wi-Fi for You ως πρωτοβουλία ε, ε, με αυτή την πρωτοβουλία μπορούν να ωφεληθούν αρχές ή ε, μονάδες ε, που, και όχι χώροι που μετά επιλέγουν τους χώρους δηλαδή ε, και το τι μπορούν ακριβώς να κάνουν. Ορίσαμε ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι ελεύθερα, να μην έχουν περιορισμούς. Οι περιορισμοί είναι η ταχύτητα και όγκος των πληροφοριών. Επίσης, Ξεσφαλίσαμε ότι οι πόροι για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι παραπληρωματικοί. Έχουμε το δέσμι της Κομισιόν, αλλά έχουμε επίσης εθνικά κονδύλια και άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ενισχύσαμε την ιδέα της ε, γεωγραφικής ισορροπίας με την έννοια της, ε, της, της καθολικότητας της όλων, δηλαδή θεωρούμε ότι κάθε χώρα στο πρόγραμμα εργασίας της μπορεί να έχει μεταβλητές επιλογές, αλλά ότι με αυτή τη γραμμή ε, ε, πλαισίωσης ενισχύσαμε την προοπτική της ε, καταπολέμησης της ε, του ψηφιακού αποκλεισμού. Επίσης, αποσαφηνίσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν φραγμοί σε σχέση με την γλώσσα ε, πρόσβασης. Ε, ορίσαμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτές οι συνδέσεις ε, στο πλαίσιο τούτης της πρωτοβουλίας θα πρέπει να έχουν μια μίνιμουμ εγγυημένη λειτουργία για τρία χρόνια, αν και η προσδοκία είναι ότι αυτοί οι σπόροι θα βλαστήσουν και θα ανθίσουν για πολύ, θα φορήσουν για πολύ περισσότερο καιρό δεν δεσμευόμαστε από κάποια τεχνολογία και εστιάσαμε όλη μας την προσέγγιση ακριβώς για αυτό το λόγο, όχι στην τεχνολογία αλλά στην ε, δυνατότητες τεχνολογικής πρόσβασης, στην γεωγραφική ισορροπία και στην ποιότητα της εμπειρίας. Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά θα μας επιτρέψουν κανονικά να επιτύχουμε και να βελτιώνουμε διαρκώς τις προβλεπόμενες ημερομηνίε έτσι, ε, έτσι ώστε επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, το έχω ήδη επαναλάβει αρκετέ φορέ, πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια αναφορά για την ανάπτυξη τη ε, σχετική συζήτηση και άρα λοιπόν όσο περισσότερο εξαπλωθεί τόσο καλύτερο και θα θέλαμε την Κομισιόν να δημιουργηθούν οι προποθέσει ώστε εντός του έτους ήδη να υπάρξουν υποψηφιότητα και συνδέσεις ήδη με το Wi-Fi for you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκιώδης τώρα. Η κυρία Γκροστέτ Εξ ονόματος κύριε Σάντερ, ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι εγώ σκιώδη για το ΕΛΚΑ, αλλά παίρνω το λόγο για, τη συνάδελφο Σάντερ που ζητά συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να φύγει νωρίτερα από ό,τι είχε προβλέψει σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεννόηση και το συμβαστικό πνεύμα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το ΕΛΚΑ στηρίζει απόλυτα την πρωτοβουλία ε, ε Wi-Fi for you. Ε, ε, και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες ε, γιατί ο κόσμος τις χρειάζεται ειδικά στις περιοχές της υπαίθρου. Κάποια θέματα ακόμα θα πρέπει να ρυθμιστούν. Πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουμε ότι το ίντερνετ θα παραμείνει δωρεάν και ανοιχτό για όλους, ενώ θα εγγυόμαστε την προστασία από τις καταχρήσεις, ιδιαίτερα για να προστατευτούν οι ανήλικοι. Ε, και έπειτα να εξασφαλίσουμε την καλή κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των χωρών, διδυρώντας στην αρχή ότι ο πρώτος που φτάνει είναι ο πρώτος που εξυπηρετείται. Η συνάδελφος Άντερ είναι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμφωνία γρήγορα ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε φυσικά να ωφεληθούν οι πολίτε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση αυτή. Κυρία Φαν από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς έχω τελείως διαφορετική γνώμη σε αυτό το φάκελο από τις συμβιβαστικές προτάσεις ε, που προέκυψαν από τις ε, άτυπες ε, ε, συναντήσεις, γιατί υπάρχουν λαϊκιστικά σχέδια εδώ αξίας 120 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι πεπισμένη ότι δεν θα πείσουν όλα αυτά ε, τον Ευρωπαίο πολίτη για την προσθέμενη αξία της Ευρώπης δίνοντας ε, δωρεάν ε, Wi-Fi. Νομίζω ότι αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα επενδύσουμε πολύ καλύτερα σε ζητήματα υποδομών για να δώσουμε πραγματική βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων εκεί όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Το Connecting Europe Facility, για παράδειγμα, έχει αποδείξει την προσθέμενη αξία του. Ε, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών και άρση στενοπών. Η πρόταση που έχουμε τώρα επιτάπητος νομίζω ότι ε, σαν άσως από το μανίκι του Γιούνκερ χωρίς ε, να υπάρχει καμία αναφορά στο πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές πόλεις και περιφέρειες ήδη παρέχουν δωρεάν ίντερνετ ασύρματο, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε και κατόπιν δημόσιας πρωτοβουλίας σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει εξολόγηση τύπου για να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα, αν υπάρχει ζήτηση ε, και πόσους πολίτες θα ε, φτάναμε έτσι είναι μια μεγάλη εκστρατεία ε, διαφημιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν έχει καμία σχέση ε, με τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο βέβαια, κανένα όφελος. Όπως το προτείνει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, τα χρήματα θα πήγαιναν σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν σύνδεση στο ίντερνετ, όμως μπορούμε να αναρωτηθούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος εάν ξαφνικά μια χούφτα άνθρωποι μόνο έχουν ε, πρόσβαση σε δωρεάν διαδίκτυο. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ε, προκλήσεις ε, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή και μπορούμε εκεί να δαπανίσουμε τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω, Πρόεδρε, ότι εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα θέλουμε να πετύχουμε σε βιβασμούς. Όμως φοβάμαι ότι για μένα αυτή η πρόταση είναι κόκκινη γραμμή και αντιβαίνει ε, σε όλες τις αρχές της χρηστή διακυβέρνησης. Δυστυχώς λοιπόν δεν θα είμαι σε θέση να την ε, στηρίξω αυτή την πρόταση με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συνάδελφος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση αυτή με βρήκε να αρχίζω διαβουλεύσεις με κάποια επιφύλαξη. Όπως είπε και ο συνάδελφος του ECR, βλέπω πως αυτή είναι μία άσκηση. Μία άσκηση για να δοθούν κινήτρα για την υπόλοιπη δεσμή μέτρων. Από την αρχή το είπα σαφώ ότι μπορώ να αναλάβω έναν επικοδομητικό ρόλο από τη στιγμή που καταλάβουμε όμω όλοι ότι η όθηση, τα ρίσματα είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να, να αλλάξουμε ε, κουλτούρα, να αλλάξουμε τρόπο μετάδοσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα αν αυτό είναι σε αστικά κέντρα ή σε περιοχές της υπαίθρου. Και σε καμία περίπτωση δεν θα δείξω προτίμηση στο μέλλον σε παράταση. Ακριβώς διότι πρέπει να είμαστε γρήγοροι για να δώσουμε αυτά τα κίνητρα. Νομίζω πως υπάρχει γενικότερα κάποια συνένεση μεταξύ του, των σχεδόν εισηγητών. Νομίζω πως έχουμε καταφέρει μια σχετική ισορροπία ε, ανάμεσα στο πώς ε, θα εξυπηρετηθούν, δηλαδή είτε σε αυτόν που έχει περισσότερη ανάγκη, είτε σε αυτόν που προλάβει πρώτος. Και νομίζω πως το κείμενο στην συμβαστική πρόταση 8 αναγράφεται αυτό όπου αναφέρεται η ισορροπία ανάμεσα στο γεωγραφικό χάσμα και το ψηφιακό χάσμα. Δηλαδή αναφερόμαστε στην Ήπεθρο και σε απομακρυσμένες περιοχές ε, όπου είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η συνδεσιμότητα. Νομίζω πως αν διαγραφεί η τελευταία πρόταση θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μετά, χρειάζεται αξιολόγηση. Εγώ θέλω να δω αυτή την αξιολόγηση και ε, feedback να... από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες βέβαια, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει επιστοποιήσει κάποιους προμηθευτές. Δεν ξέρω ακριβώ τις λεπτομέρειες, αλλά θα γίνει μια αξιολόγηση όχι μόνο για τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί σε συγκεκριμένα έργα, αλλά για να δουν αν έχει αυτό ε, το... αυτές τις ε, πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα σε εμά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί νομίζω πως Εάν καταφέρουμε τις συνέργειες, τότε και θα προάγουμε τη συνδεσιμότητα και ε, θα δίνει μία περιοχή την όθηση στην άλλη για να ε, επιταχύνει τις προσπάθειες σύνδεσης. Παρά λοιπόν την αρχική μου επιφύλαξη, συντομεύεται λέει ο Πρόεδρος, παρά την αρχική μου λοιπόν επιφύλαξη, νομίζω πως οι συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες καταλήξαμε είναι τροπολογίες που μπορώ να εγκρίνω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ηλικιώτη από την ΚΟΥ έχει το λόγο τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Κάρλο Ζωρίνιο για την παραγωγική συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση των εισηγητών και δι για την προσπάθεια του να λάβει υπόψη τι προτεραιότητε όλων των πολιτικών ομάδων. Συμφωνούμε με τη θέση του εισηγητή πω πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει δωρεά διασύνδεση υψηλή ποιότητα σε χώρου όπου παρέχονται δημόσιε υπηρεσίε και χαιρετίζω με την πρότασή του να συμπεριλάβει στου συμβαστικέ τροπολογίε και του επιπλέον τόπου όπου έχουμε προτείνει για να υπάρχει δωρεά διασύνδεση όπω είναι τα πανεπιστήμια, οι χώροι δημόσιων συγκοινωνιών καθώ και άλλου χώρου κοινωνική ζωή. Επίση, συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί πω ο διαθέσιμο προπολογισμό θα κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο και να στηριχτούν ιδιαίτερα τα κράτη και οι περιοχέ που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, η θέση αυτή αναιρείται από την πρόταση πω ο προπολογισμό πρέπει να κατατίθεται κατά κανόνα με βάση τη σειρά παραλαβή των προτάσεων. First come, first serve. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν δυο λογικέ που είναι αντίθετε. Γι' αυτό επιμένουμε πώ πρέπει να διαγραφεί αυτή η αναφορά το first come, first serve και αντί αυτού να προσθεθεί πω πρέπει να στηριχτούν επαρκώ τα κράτη και οι τοπικέ αρχέ ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τι προεργασίε για την υποβολή αιτήσεων. Για την ομάδα μα είναι προτεραιότητα να αποφερθούν από την ασύρματη συνδεσιμότητα ιδιαίτερα τα κράτη και περιοχέ που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε, τα νησιά, οι ορεινέ παραμεθόριε, οι απομακρυσμένε και οι δυσπρόσιτες περιοχέ. Στόχο μα είναι να εξυπηρετούν οι ανάγκε όλων των πολιτών, να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό δημόσιο όφελο και να δοθεί η δυνατότητα στου πολίτε από όλα τα κοινωνικά στρώματα να επιφορηθούν από τα πλεονεκτήματα τη συνδεσιμότητα. Τέλο, θεωρούμε πω πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα πω η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ω δωρεάν μόνο εφόσον παρέχεται χωρί χρέωση, είτε αυτή γίνεται υπό τη μορφή άμεση πληρωμή, είτε έναντι άλλου τμήματο, συμπεριλαμβανομένη μεταξύ άλλων τη διαφήμιση και τη παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι τροπολογίε που ε, έχουμε καταθέσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε.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 Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην εφαρμογή να αναζητηθούν ε, συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια και να είναι εγγυημένη η ένταξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών ή σε μετάβαση ώστε να εγγυηθούμε την κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης ε, στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος. Ε, Επίσης πρέπει να εισηχθούν εγγύησεις ε, για τις ελάχιστες προδιαγραφές υψηλής ε, ταχύτητας ε, ή της μέγιστης ταχύτητας που υπάρχει στην αγορά. Ευχαριστώ. Oh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Connect. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε και εμείς τη σύγκληση και τη συμφωνία, τη σύγκληση απόψεων ανάμεσα στα μέλη αυτής της Επιτροπής. Η κύρια ανησυχία μας ε, αφορά το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ανέφερε και ο εισηγητής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και μας χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι εδώ στο Κοινοβούλιο ε, δουλεύεται πάρα πολύ γρήγορα. Αναφέρθηκαν ανησυχίες ε, σχετικά με τον προπολογισμό. Αυτό χρειάζεται προσοχή για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια γρήγορη συμφωνία στον τριμερή διάλογο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπόλοιπες διαστάσεις που αναφέρθηκαν, οι περιορισμοί στην νομοθεσία αναφέρθηκε πως θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και πως θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους τύπους ε, κοινοτήτων, πόλεων, υπαίθρου κτλ. Και να μην ε, υπάρχει έλλειψη ισορροπίας. Και εμάς μας ανησυχεί το ίδιο όσο και εσάς, ιδιαίτερα στο στάδιο της εφαρμογής. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε αυτά τα κουπόνια να τα διανύμουμε ε, ίσα σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Επίσης θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες συμπληρωματικέ μεθόδους χρηματοδότησης, ταμεία κτλ. Και η πρακτική Εκεί που έχουμε προτείνει, το First Call, ε, συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, χρηστή διαχείριση, τακτική υποβολή εκθέσεων, έτσι ώστε να πετύχει το εγχείρημα αυτό σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Ζωρίνιο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις συμβολές τους. Το θέμα του προπολογισμού σίγουρα θα είναι θέμα κλειδί στο τριμερί. Σε αυτή την φάση, το που θα, αν τεθεί στο επιτάπητο θα είναι από την ε, Επιτροπή Προπολογισμού, αλλά βεβαίως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας βρει ενωμένους ε, να δουλέψουμε με ε, σταθερό τρόπο. Έχουμε 25 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα. Και επιπλέον θα πρέπει να συνδυάσουμε, όπω είπαμε, εθνικά κονδύλια και κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία. Από την άλλη πλευρά είναι μια προσπάθεια που κάνουμε. Προσπαθούμε να, να φτιάξουμε καλύτερε συνθήκες, ιδιαίτερα για τα θέματα που τίθενται στον ορισμό του τι πρέπει να είναι, ε, τι πρέπει να είναι οι ορισμοί, οι περιορισμοί μάλλον, καθολικότητα για όλου. τον, έφερε και ο συνάδελφος Ηλικιώτη και ακριβώς το έχουμε να πει ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η πτυχή. Η παρακολούθηση επίσης και αυτή έχει τεθεί επανειλημμένα. Προσπαθούμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ε, εξάπλωση ε, αλλά και στον χρονισμό γιατί τα εθνικά προγράμματα είναι αυτά τα οποία θα συσπίζουν τα κριτήρια που διασταυρώνουν αυτή τη λογική του first come, first served, δηλαδή όποιος φτάσει πρώτος εξυπηρετείται πρώτος και πρέπει εκεί να βρούμε μια ισορροπία και όντω αυτό να ζητούμε Πρόεδρε, ε, σωστή ισορροπία και σε σχέση με τα όσα είπε η συνάδελφος του ECR, όπως είπε και πολύ ξεκάθαρα η ίδια θεωρεί μάλλον η ομάδα, η e θεωρεί ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι ε, πόροι που να είναι καλύτεροι. Εμείς δεν το ε, θεωρούμε αυτό. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα ώστε να εκμεταλλευτούμε τους πόρους που προβλέπονται από αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Ε, αυτά. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Να θυμίσω, είναι βέβαια γραμμένο και στους φακέλους σας ότι έχουμε ψηφοφορία στις 25 Απριλίου στην Ήτρε, στην Ολομέλεια θα δούμε πότε, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά Σκιώδης και πάμε στο 18 που είναι η μελέτη με θέμα την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογή σχετικά με το Horizon 2020. Έχουμε τους ερευνητέ μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, την, Υπηρεσία ερεύνηση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το EPRS. Α, είστε εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, φτάνει και ο κύριος Διευθυντής. Σε ένα λεπτό. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Μόνο γιατί είναι και η δική μου ε, μας έκθεση για την εφαρμογή του Horizon 2020. Τον το επόμενο μας θέμα είναι η Soledad Capeson Ruiz, είναι η συγχύτρια. Και ε, γι' αυτό και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα εσείς πιστεύετε για τη δική μας αξιολόγηση. Κατάλαβα ότι αυτή είναι, αυτό είναι το βασικό ζήτημα που θα αναφέρετε από δική σας πλευρά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάκο είναι από την Υπηρεσία Ερευνών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα θέλω να επισημάνω ότι αυτή η αξιολόγηση ε, του προγράμματος Horizon 2020 ε, αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος ε, αξιολογήσεων υλοποίησης που υπάρχει τις θερμοδιότητες της, ε, της Υπηρεσίας ε, Ερευνών του Κοινοβουλίου. Θα σταθώ στις τρεις προτεραιότητες του προγράμματος Horizon 2020 από πλευράς έρευνας και βιομηχανίας και ο συνάδελφος θα εξετάσει άλλες πτυχές. Πρώτα απ' όλα, ε, στις εξαιρετικές προτεραιότητες τις ερευνητικές είδαμε ότι υπάρχει ευρύτατη και ισχυρότατη στήριξη σε όλη την Ευρώπη για αυτό το τμήμα του προγράμματος. Με την πεποίθηση ότι συμβάλλει σημαντικά στην ερευνητική αριστεία ε, και ανταγωνιστικότητα στην έρευνα και την καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο έχει ισχυρότατη στήριξη και είναι μια πραγματική ιστορία επιτυχίας. Οι ε, δομές ε, ερευνητικής βιομηχανίας έχουν συμβάλει ιδιαίτερως ότι αφορά την ε, επιτυχή ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υποδομών. Οι μελλοντικέ τεχνολογίες έχουν συμβάλει σημαντικά στην ηγετική θέση της Ευρώπης σε τομείς όπως είναι οι κρατικέ τηλεπικοινωνίες, τα nanoelectronics και ε, προηγουμένη ρομποτική. Και με τις δράσεις μας έχουμε προσελκύσει διεθνές ε, ταλέντο στην Ευρώπη ε, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την βιομηχανική ηγεσία, βλέπουμε ότι η βιομηχανία Εκτιμώ ιδιαίτερω ε, την αύξηση της χρηματοδότησης για τις γενοτόμε δράσεις, ιδίω ε, τα νέα μέσα για τις μικρομεσαίε επιχειρήσει και το Fast Track Innovation, καθώς και την ενισχυμένη χρήση των εργαλείων ε, με γνώμονα την βιομηχανία, όπω είναι οι συμπράξει δημοσίου τομέα. Η μειωμένη χρηματοδότηση για την θεμελιώδη βασική έρευνα έχει δυσμενείς επιπτώσεις ε, για τα ερευνητικά ιδρύματα και εντοπίσαμε ότι η συνεργασία μεταξύ έρευνα και βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό μένει στα μέσα επίπεδα TRL. Σε συγκεκριμένες τεχνολογίες σχεδόν 52% των επιδοτήσεων αφορούν ε, επιχειρηματικές ε, ενώσεις παρότι συνήθω είναι μικρές, 26,7% ε, των συνολικών συνεισφορών. Σε αυτόν τον τομέα πιο συγκεκριμένα, ε, σε ό,τι αφορά την ε, τεχνολογία της πληροφορικής, η γενική προσέγγιση θεωρείται ικανοποιητική σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, όπως είναι τα μαζικά δεδομένα, υπολογιστική ισχύ, το διαδίκτυο των αντικειμένων και βασικά ευρήματα τώρα για τις κοινωνικές προκλήσεις. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ προκλήσεων στη συμμετοχή ε, των ε, κερδοσκοπικών ε, επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στις μεταφορές, 55,3% της συμμετοχής αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ στην... αλλά και μάλλον και στη τομέα της ενέργειας, ενώ στην, στον τομέα της υγείας, της δημογραφικής αλλαγής και της ευημερίας μόνο 27,2% και στον τομέα Ευρώπης, σε έναν ε, κόσμο που αλλάζει είναι μόλις 17,9%. Βλέπουμε λοιπόν όλες αυτές τις διαφορές που εν μέρει εξηγούνται από τις εγγενείς ε, διαφορές. Έχουμε την ανάγκη για βασική έρευνα σε επιμέρους τομείς. Όμως, Υπάρχει και μια επιλογή εργαλείων σε αυτούς τους τομείς ε, που ε, οδηγεί τη συμμετοχή προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες ε, δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα, όπως είναι η πρωτοβουλία καινοτόμων φαρμάκων. Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες. Εξετάζοντα τα συνολικά, θεωρήσαμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν υπόψη. Πρώτον, οι πολύ ανταγωνιστικέ διαδικασίε επιλογή οδηγεί στη συγκέντρωση τη χρηματοδότηση σε, ε, ε, ιδρύματα αριστεία και αυτό μπορεί να αποθαρρύνει την ευρύτερη συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων του ορισμού 2020. επίση το γραμμικό μοντέλο καινοτομία, το οποίο είναι εγγενέ σε, σε πολλές διαδικασίες του Ορισμού 2020, θεωρείται μειονέκτημα ε, για τους ε, φορείς και περιφέρειες ε, έρευνας και καινοτομίας και βιομηχανίας, χαμηλής ικανότητας όμως. Πολλά σχόλια αφορούσαν τη διαρροή εγκεφάλων, όπως αποκαλείται το brain drain, που αποτελεί σημαντική πρόκληση πλέον για πολλές χώρες. Πίσω από όλα αυτά, εάν η Ευρώπη θέλει να πετύχει τον στόχο του 3% του ΑΕΠ, το οποίο θα επενδύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, τότε πρέπει κατά κάποιον τρόπο, με κάποιον τρόπο μόνο να βρεθούν ένα εκατομμύριο ακόμα νέοι ερευνητές. Η συμμετοχή στη, οι συμμετέχοντες στη βιομηχανία και έρευνα εκτιμούν τις ε, διεθνικές εταιρικές σχέσεις, θεωρούν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων, όμως η διαχείριση των μεγάλων συμπράξεων είναι και πάλι ακόμα μάλλον επαχθής. Οι συμμετέχοντες ε, θέλουν την απλούστευση, βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή τη δικασία και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ιδίως σε αφορά τον υπολογισμό του εσωτερικού κόστους και το IPR τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή εμπειριών στο πρόγραμμα, θεωρούμε ότι μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή τη βιομηχανία και ε, θεωρούν ότι το πρόγραμμα δεν φτάνει, δεν αγγίζει τις πολύ δυναμικές και καινοτόμες ε, νεοφυείς επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τέτοια χρηματοδοτικά μέσα για να ε, συνεχίσουν. Συνέργειες μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων έχουν μόλις ξεκινήσει και δεν ε, μπορούμε ακόμα να σχολιάσουμε τα αποτελέσματά τους γιατί δεν, έχουμε, δεν τα έχουμε λάβει ακόμα. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν και πτυχές ε, του ΕΦΣΥ, τα οποία και πιο συγκεκριμένα εδώ αναφερόμαστε στην ΕΦΗ e, εξειδίκευση, που δεν ε, αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ευρύτερες ε, κοινωνιακές αλλαγές, προκλήσεις μάλλον. Πρέπει να υπάρξει μια συμφιλίωση μεταξύ των μικρών και μεγάλων τέτοιων προκλήσεων. Τώρα, ως προς τις συστάσεις. Ε, πρέπει να λάβουμε καλύτερα υπόψη τις διαστάσεις των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, καλύτερη αλληλεπίδραση και άντληση διδαγμάτων σε ό,τι αφορά τις κοινωνιακές προκλήσεις, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες και απαιτείται πρόοδο ό,τι αφορά την ολοκλήρωση ε, των στοιχείων, των ανθρωπιστικών επιθυμών στην ε, έρευνα και καινοτομία. αλλά και στον τομέα της πληροφορικής. Ε, ακόμα απαιτείται πρόοδος ε, ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα μαζικά δεδομένα. Επίσης, εδώ μπορούμε να πούμε ότι τα πάνελ αξιολόγησης, ιδίως για τα υψηλά επίπεδα ετοιμότητα, τεχνολογικής ετοιμότητας, μπορούν να είναι πιο ισορπημένα σε ό,τι αφορά την σύνθεσή τους ε, με μεγαλύτερη εκπροσώπηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μας δώσατε εσείς ε, την ε, πλευρά της ε, έρευνας και βιομηχανίας. Τώρα θα περάσουμε στην οικονομία και, τα, και τη χρηματοδότηση του προγράμματος Horizon 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα, αυτή είναι μια εξελόγηση του Horizon 2020 από οικονομική χρηματοδότηση πιστοτική σκοπιά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια καλή παρουσίαση και να σας ε, παρουσιάσω τη μεθοδολογία και τις συστάσεις που έχουμε αναπτύξει. Στη μεθοδολογία έχουμε δει τα διαφορετικά εργαλεία, δεδομένα, βάσει δεδομένων που συλλέγουμε δεδομένα από όλα τα προγράμματα της Ένωσης, έχουμε δει τα ίδια τα προγράμματα που είναι στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και βασίσαμε την ανάλυση μας ε, σε συνετεύξεις, σε case studies και ε, τα λοιπά. Η αξιολόγηση είναι, αφορά τα ψηλά επίπεδα, αλλά είναι βασισμένη σε γεγονότα σε, που μπορούν ε, να, διασταυρωθούν και οι πληροφορίες που δεν θεωρήσαμε σημαντικές δεν συμπεριλήφθηκαν στις, ε, στο τελικό, στην τελική μελέτη. Καταρχάς, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν, μια, έχουν ένα καλό όραμα, έχουν ε, επίγνωση του τι συμβαίνει, είναι ενήμεροι, δεν φαίνεται στη διαφάνεια, αλλά βρίσκεται στη μελέτη. Τώρα, ένας από τους στόχους του ορίζοντα είναι να βελτιωθεί απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Επίσης αυτή ήταν και μία πολύ σημαντική έτσι που έπρεπε να απαντήσουμε στη μελέτη. Οι διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς ανέφεραν ότι είναι πολύ δύσκολο μέτρο και δύσκολο να αξιολογηθεί για διάφορους λόγους. Ε, επειδή, για παράδειγμα, κάποιες επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες, κάποιες ε, θα φανούν σε πάνω από 10 χρόνια και κάποιες, από κάποιες επιπτώσεις μπορούν να πάρουν τη μορφή καινοτομίας. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Υπάρχει ένας ε, αριθμός δικτών και στοιχείων μέτρησης, για παράδειγμα συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημοσιεύσεις κτλ. που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά ήταν πολύ γενικός και δεν ε, έμπαινε σε λεπτομέρειες τα επιμέρους στοιχεία των προγραμμάτων. Τώρα υπάρχουν συνδέσεις ανάμεσα στα προγράμματα, αλλά πρώτα ας περάσω στο σημείο 3. Διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα έπρεπε να είναι τα προγράμματα. Ορισμένοι θεωρούν ότι τα προγράμματα αυτά, έτσι όπως είναι σχεδιασμένα, θα ε, δώσουν περισσότερη βαρύτητα σε ορισμένε βιομηχανίε από άλλες. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα. Άλλοι θεωρούν πως πρέπει να υπάρχει διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στις βιομηχανίες μεγάλου κύκλου ζωής και στις ε, βιομηχανίες που έχουν μικρό κύκλο ζωής. Πώς όμως καταφέραμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και στις ε, επιφυλάξεις των διάφορων φορέων, ε, δημιουργώντας προτεραιότητες, στρατηγικές προτεραιότητες. Πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι στρατηγικές προτεραιότητες. Στόχοι του προγράμματος θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί σε, βασισμένοι στο τι μπορεί να φέρει στην κοινωνία το κάθε πρόγραμμα. Αυτό αναφέρεται σε σαφέστατα στην εκτίμηση αντικτύπου για το νωρίς το 2020. Αλλά είδαμε ότι υπάρχει μια καλύτερη διασύνθεση ανάμεσα στις προτεραιότητες και στις αιτίες και στην αγορά. Μετά, πολύ σημαντικέ είναι και οι εξωτερικές επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν αυτά τα προγράμματα και ο αντίκτυπος που θα έχει σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας. Είδαμε πως σε ορισμένα κομμάτια του προγράμματος υπήρξαν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για το ίδιο το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει υψηλή συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας που αυτό είναι θετικό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι ερευνητές συμμετείχαν, ήταν ενημερωμένοι, ήθελαν να αποτελέσουν μέρος του προγράμματος. Από την άλλη θα είχαμε πρόβλημα εάν υπήρχε χαμηλή συμμετοχή και εάν ορισμένα κομμάτια του προγράμματος ε, είχαν ελάχιστους συμμετέχοντες. Ωστόσο, Υπάρχουν και οι αρνητικές επιπτώσεις. Μας είπαν, για παράδειγμα, ότι ορισμένοι συμμετέχοντες κοίταξαν τα ποσοστά επιτυχίας προτού κάνουν αίτηση για τα διάφορα προγράμματα. Και αυτό σίγουρα έχει άμεσες επιπτώσεις ε, γιατί δεν θα γίνονται αιτήσει για κάποια προγράμματα. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι οι ερευνητές να αντιμετωπίζουν το πρόγραμμα αντικειμενικά. Και αυτό θα έχει αμέσως επιπτώσει στη διαδικασία αξιολόγηση των των διαδικασιών υποβολής προσφορών. Είναι πολύ βασικό όλο το πρόγραμμα να βασίζεται στην ομιμότητα της αξιολόγησης μιας πρότασης. Επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη διαφάνειας και να αξιολογήσουμε τα προσόντα που έχουν όσοι θα κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Μετά έγινε σημαντική πρόοδος στη διαδικασία αξιολόγησης και στην απλοποίηση. Ε, είδαμε ότι η απλοποίηση έχει κάποια προτίμηση σε έγκριτους ερευνητές, σε ήδη καθιερωμένους ερευνητές και σε συγκεκριμένες ε, εταιρείε που βοηθούν για να δοθούν επιχορηγήσεις. Μετά, είδαμε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση κονδυλίων σε ορισμένους. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, να μιλάτε πιο αργά. Το ξέρω. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν, νομίζουμε, πολλοί στόχοι και μπερδευόμαστε. Από τη μία θέλουμε δηλαδή εξαιρετική επιστήμη, θέλουμε αριστεία, από την άλλη θέλουμε τα πάντα για την κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό που οδηγούμαστε στις συστάσεις. Καταρχάς, ε, πρέπει να ορίσουμε το πρόβλημα, πρέπει να ορίσουμε τους διαφορετικούς ε, στόχους. Αυτό χρειάζεται όχι μόνο έναν καλύτερο ορισμό που έχει διγίνει, αλλά και καλύτερη επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μετά θα μπορούσε να γίνει μία ε, εκ νέου αξιολόγηση του σχεδιασμού της αγοράς και ε, το γιατί υπάρχουν προγράμματα που έχουν αποτύχει. Θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να αξιολογήσουμε γιατί υπήρξαν αυτές οι αποτυχίες στην αγορά, πώς και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει και στη διεξαγωγή των ελέγχων και στην, στον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων, έτσι ώστε να αποφύγουμε να επαναλάβουμε τα πιο κοινά λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας μένει χρόνος, δυστυχώς, και επιτρέψτε μου, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ότι αυτοί οι τρεις κύριοι που έχουμε καλέσει, δύο ερευνητέ και ο Γενικός Διευθυντής Ρομπέρτ Γιάννη Σμιθ θα είναι εδώ και όταν θα συζητήσουμε την αξιολόγηση εφαρμογή για το ορίζοντα 2020, για το επόμενο δηλαδή σημείο της ημέρησης διάταξης. Γι' αυτό, αν έχετε κάποιες σύντομες ερωτήσεις προς τους προσκεκλημένους μας, θα έχετε τη δυνατότητα να τις κάνετε. Έχουμε την εξαιρετική αυτή ευκαιρία. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε, να τους εκμεταλλευτούμε, αλλά και όταν θα έχει τελειώσει η συνεδρίαση, γιατί βλέπω πως δεν μας μένει πολύς χρόνος. Αν έχετε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις, έχετε τη δυνατότητα να τις κάνετε τώρα. Κυρία Νίμπλερ, θέλετε τώρα να κάνετε την ερώτησή σας. Α, θα περιμένετε αργότερα. Τέλεια. Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στην έκθεση. Η συγγήτρια είναι η Σολεδάδ Καπεζόν. Είστε έμπειροι, ξέρετε πολλά για αυτό το θέμα και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να μπορέσουμε όντως να συζητήσουμε και να ακούσουμε σχόλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η πρόταση έκθεσης έχει ως στόχο να εξισορροπήσει όλα τα συμφέροντα και τις απόψεις. Γι' αυτό Έχουμε το τρίγωνο της επιστήμης, των πανεπιστημίων και της εμπειρίας και εμείς βλέπουμε ότι ε, έχουμε μια πολύ σκόπιμη αξιολόγηση εφαρμογής σχετικά με το ρίζοντας 2020 και έχουμε επίσης και αποστολές που κάναμε εγώ ε, και οι συνάδελφοι στην Πολωνία, στην Ισπανία, ε, στην Πορτογαλία για να δούμε από πρώτο χέρι πώς κατανέμονται αυτά τα χρήματα, πώς γίνεται η συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αν ήταν επιτυχές αυτό το πρόγραμμα. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσω με μια αξιολόγηση πολύ θετική που δεν προαπορεί μόνο από μένα την ίδια, αλλά από όλους τους συμμετέχοντες που ε, μετέβησαν ε, επί τόπου. Η αξιολόγηση είναι πολύ θετική λοιπόν και ε, γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω ενίσχυση του πρωτοβουλία αυτής. Ε, επίσης, η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα είναι σημαντική για το επόμενο πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο. Τέταρτον, και έτσι ολοκληρώνω και τις γενικές μου παρατηρήσεις, ότι το θέμα της αριστείας θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα και στο επόμενο πρόγραμμα ε, μέχρι το 2020, το οποίο προκύπτει μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης, όπου η ανάγκη καινοτομίας έχει σηματοδοτήσει όλη αυτή την περίοδο. Τώρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέοι στόχοι που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το μέλλον. Ε, όπω ξέρουμε υπάρχει το πρόβλημα του λαϊκισμού, της ασφάλειας, της θερμοκρατίας, της ξενοφοβία. Και τώρα για συγκεκριμένα σημεία θέλω να αναφερθώ από το οικονομικό ζήτημα, από το προπολογισμό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μεγάλη μεγάλη μεγάλη επιτυχίες ε, λόγω της μεγάλη συμμετοχής και των αριθμών αριθμό των project, των πολύ σημαντικών project, αλλά δυστυχώ μόνο το 14% πετυχαίνει τη χρηματοδότηση και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μεγάλο κομμάτι των project που δεν χρηματοδοτούνται είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτό με μια ε, αναλογία 1 στα 11 δηλαδή προγράμματα εγκρίνονται και αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για σημαντική αύξηση του 8ου προγράμματος και χρειάζεται όμως μεγαλύτερη προσπάθεια για το επόμενο ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Ένα δις ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα, είναι το σημαντικότερο στον κόσμο της έρευνας. Δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, δεν μπορεί να είναι το μόνο πρόγραμμα που επιτρέπει αυτή την ανταγωνιστικότητα και την αριστεία στην Ευρώπη που θέλουμε. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια όλων των χωρών, όλων των φορέων, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το 3% όπου έχει καταλήξει ε, το Συμβούλιο της Βαρκελόνης. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια προσπάθεια από όλες τις αλλά και από την ίδια τη βιομηχανία. Ο ιδιωτικός τομέας καταβάλει σημαντική προσπάθεια αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα ώστε να μπορέσει και εκείνη να συμβάλλει κατά τα δύο τρίτα που πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί 70 με 90% είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη κυρία μου. Μάλλον πρέπει να διαβάσετε λίγο αργότερα, ε, λίγο πιο σιγά, γιατί οι διερμηνείς μας ε, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την ταχύτητα. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε όλα όσα λέτε. Χάνετε, χάνετε το νόημα αν διαβάζετε με τέτοια ταχύτητα. Μάλιστα, συνεχίζω και θα διαβάσω λίγο πιο αργά. Έρευνα λοιπόν ε, και καινοτομία από και για την κοινωνία. Το πρόγραμμα ορίζοντα 2020 θα πρέπει να δώσει απαντήσει στους διαφορούς στόχου, και ζητάμε να υπάρχει εγγύηση απόδοσης προς το κοινό, ώστε δηλαδή να μην δημιουργούνται νέε ανισότητες, ιδιαίτερα στις ευαίσθητε περιοχές, ε, περιφέρειε. Πρέπει να δοθεί επίσης ένα συγκεκριμένο μήνυμα με την επιστημονική διπλωματία, ιδιαίτερα με τις κοινωνικές εξελίξεις. Λυπούμεθα γιατί ένα 5% Πέρασε μόνο στο 8% η συνεργασία η αναπτυξιακή. Ε, και όσον αφορά την επιστημονική συνεργασία και τη συνεργασία των κέντρων αριστείας. Χρειαζόμαστε περισσότερα κέντρα αριστείας και περισσότερες περιφέρειες αριστείας. Χρειαζόμαστε λοιπόν να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ περισσότερων κέντρων αριστείας η συγκέντρωση εγκεφέλων θα πρέπει να αποφεύγεται και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των λόγω κέντρων αριστείας στην έρευνα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι ως συμπέρασμα, λέει ο Πρόεδρος. Ναι. Συντονισμό, συνεργασία λοιπόν και η μελέτη του Πιερές λέει ότι δεν υπάρχει χρόνος, ότι, μάλλον χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Εγώ πιστεύω πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός. Τα διευθυντικά ταμεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ε, ε, και εκεί προγράμματα και την αρχή της παραπληρωματικότητας και της συμβατότητας ανάμεσα στις ρυθμίσεις και για τα φύλλο έχουμε φτάσει το 50% όσον αφορά τη συμβουλευτική εργασία αλλά εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο 40% εμπειρογνωμόνων γυναικών στα πάνελ και στα project. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το θέμα του φύλλου όταν αξιολογείτε το κάθε project. Θα πρέπει λοιπόν τα αποτελέσματα να εφαρμόζονται. Ε, ναι, ναι, και κλείνω. Αξιολόγηση αριστεία όπως είπα χρειάζεται να ορίσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο, περισσότερη διαφάνεια και να έχουμε κριτήρια κοινωνικά και φύλου. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τα ποσοστά των όσων έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχουν και περιοχές όπου δεν έχει γίνει κανένα πρόγραμμα και όσον αφορά τη μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος των συμμετεχόντων και του ε, κλάδου κάθε φορά, εγώ θεωρώ πως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο ε, ξεκάθαρα, γιατί υπάρχει προστεθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, θα μπορείτε να προσθέσετε κάτι στο τέλος ε, της συζήτησης ως συζητήτρια που είστε συνοψίζοντας ίσως λίγο, γιατί τώρα πρέπει να περάσουμε και να ακούσουμε τους σκιώδες εισηγητές. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά αν από τα μέλη μας, η κυρία Αγγέλικα Νίμπλερ από την αρχή ήθελε να πει δύο λόγια και να ρωτήσει κάτι και μετά θα περάσουμε στους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την ειλικρινή ανοιχτή διαφανή τους ανάλυση. Ο ορίζοντας 2020 είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πολύ που είμαστε τόσο ανοιχτοί. Είδαμε λοιπόν μετά από την ανάλυση αυτή που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχει ανάγκη να γίνουν διορθώσεις και θα ήθελα αυτό να το πω ευθύ εξ αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Συνήθω κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως δεν είναι ανοιχτή στο διάλογο, αλλά αυτή τη φορά αποδείξατε το αντίθετο. Ε, τώρα, αν έχω καταλάβει καλά, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στο δρόμο της καινοτομίας. Απομακρυνθήκαμε κάπως από αυτό, έτσι ώστε να δημιουργηθεί περισσότερη... Ε, να γίνουν πιο ελκυστικά τα προγράμματα, να έχουμε περισσότερες αιτήσει από ενδιαφερόμενους, από ερευνητέ κτλ. Είδαμε πως υπάρχει μια συγκέντρωση ε, στου, σε συγκεκριμένα πράγματα, σε δημόσιους διαγωνισμούς, υπάρχει έλλειψη ε, κινήτρων, αλλά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε και νομίζω πως εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση, να ξαναδώσουμε βάρος στον ίσο, ε, στην ίση κατανομή των ε, αιτήσεων για έρευνα και να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους για να μπορούμε και να τους επιτύχουμε. Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους, διακόπτει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οι σκιώδες τώρα. Κυρία Κουτρίτσκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά νόμιζα ότι η Αντζέλικα είναι σκιώδης συγχυτριά μας, γιατί σχολίασε τα όσα υπόθηκαν ε, απευθείας. Θα υπάρξει και συζήτηση βέβαια στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σολεδάδ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Πραγματικά κατέβαλε σημαντικέ προσπάθειε σε αυτήν την έκθεση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο. Όμως σε συγχαίρω για τη δουλειά που έχεις κάνει. Οι συστάσεις μας, εδώ είναι το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά το ένα, το πρόγραμμα πλαίσιο. Σε πολλές συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε αποστολές στην Ισπανία, στην Πορτοκαλία, Γερμανία, Πολωνία, είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συναντήσουμε επιστήμονες και εκπροσώπους της βιομηχανίας. Και ακούσαμε λοιπόν τα προβλήματα, τα σχόλιά τους. Συμφωνούμε με πολλές από τις προτάσεις. Πράγματι και ο περιπολογισμός του επόμενου προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να αυξηθεί στα 100 δις ευρώ. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο η δομή των τριών πυλώνων, όμως ο τρίτος πυλώνας κοινωνιακής ε, προκλήσης θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος. Βέβαια, εμείς θα ζητήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ του ένα του προγράμματος πλαισίου και των διαρθρωτικών ταμείων. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ικανών των κρατικών ενισχύσεων με το κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη και χρειάζεται απλούστευση και σαφήνεια σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ιδίως σε σχέση με την ε, δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομία. Σημαντικό επίσης είναι αυτό που ανέφερε η Σολεδάδο, ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία στη χρηματοδότηση έρευνα και καινοτομία, καθώ και μεγάλων και μικρών έργων να βελτιώσουμε την συνεργατική έρευνα, όπως είπε και η Σολεδά, και κάτι άλλο σημαντικό, και το συζητήσαμε κατά τις συναντήσεις μας, ότι για η χρηματοδότηση για ε, την αμυντική έρευνα θα πρέπει να είναι εκτός του ένα του προγράμματος πλαισίου και η Επιτροπή ήδη ακολουθεί αυτή την άγουσα. Στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να αντισταθμίσουμε αυτό το πλεόνασμα αιτήσεων ε, που τελικά οδηγεί σε πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Δεν έχουμε εδώ συγκεκριμένες προτάσεις, όμως αυτός θα πρέπει να είναι ο σκοπός του ένα του προγράμματος πλαισίου. Αλλά και η διεύρυνση της συμμετοχής. Ε, πάντα το λέγαμε αυτό, δεν είναι κάτι το καινούριο. Αλλά να έχουμε και περισσότερα μέσα για την διεύρυνση της συμμετοχής, αλλά και περισσότερες ε, δαπάνες, περισσότερα κονδύλια. Τέλος, ε, τα ζητήματα των γυναικών. Το αναφέρατε προηγουμένως. Συμφωνώ ότι είναι λίγες ε, οι γυναίκες που εργάζονται στα πάνελ αξιολόγησης των αιτήσεων. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διορθώσω αυτή την κατάσταση. Όμως δεν συμφωνώ με την πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα επιπρόσθετο κριτήριο ε, προτιμησιακής αντιμετώπισης, αν θέλετε, για τις γυναίκες ε, επιστήμονες. Εγώ δεν ε, συμφωνώ. Ακόμα και οι πλέον φεμινίστριες των επιστημόνων δεν θα υποστήριζαν κάτι τέτοιο ένα τέτοιο κριτήριο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι είναι πιο αδύναμες από τους ε, άνδρες επιστήμονες και χρειάζονται ε, κάποιο άλλο πλεονέκτημα για να τους ανταγωνιστούν. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι με βάση την αριστεία, όχι με άλλες ε, προτεραιότητες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στο πάνελ εξελόγηση δεν θα πρέπει να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Πρέπει να σημαίνει κάτι τέτοιο. Κλείνοντας να ευχαριστήσω τον κύριο Έγκερτ για τη συνεργασία του. Όταν, ε, κατά την προετοιμασία των ε, παρατηρήσεων, ευχαριστώ όλους τους χιώδεις. Ήταν πολύ ενεργός η συμμετοχή όλων. Ευχαριστώ από πλευρά CCR. Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι πολύ ικανοποιητικό η έκθεση της συζητήρια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αντανάκλαση των συζητήσεων που έχουμε κάνει ήδη στις συναντήσεις ε, των σκιωδών και βάσει των επισκέψεων που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της έκθεσης. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον την Επιτροπή Ερευνών του Κοινοβουλίου, γιατί νομίζω ότι μας έδωσε πολύτιμες ε, πληροφορίες ε, και στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας ορίζουν 2020 που έχουμε στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ορισμένα ζητήματα κρίσιμη σημασία για μένα. Πρώτον, και έχει ήδη αναφερθεί, πρέπει να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το Brexit. Δεν θέλουμε να αυξηθεί γενικά ο προπολογισμό. Ε, να είναι πιο ε, φιλικό προς τις επιχειρήσεις το πρόγραμμα σε σχέση με το ορίζον 2020. Βλέπουμε ότι για τις επιχειρήσεις είναι ακόμα πολύ δύσκολο να ε, συμμετάσχουν σε ένα έργο υπό το ορίζον 2020. Υπάρχει διοικητικό άκτος το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δίνεται μεγαλύτερη ανατροφοδότηση μετά την απόρριψη ενός έργου και Νομίζω ότι έτσι μαθαίνουν και οι αιτούντες ε, κάτι παραπάνω, αντί να νιώθουν απλώς ε, θυμό και αγανάκτηση και απογοήτευση. Ε, πρέπει να έχουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα κονδύλια και ένας τρόπος είναι να έχουμε consultants, όμως περισσότερα χρήματα πάνε προς αυτούς τους συμβούλους παρά προς τα ίδια τα έργα τελικά. Αυτό είναι το πρόβλημα το πρώτο βήμα αξιολόγηση είναι σημαντικό γιατί έτσι αυξάνεται ε, σημαντικά ίσως ε, το ποσοστό συμμετοχής ε, και επιτυχίας. Κάποιες φορές πρόκειται και για σπατάλη χρημάτων και ενεργειών για τις επιχειρήσεις, το να μην περάσουν στο δεύτερο στάδιο. Ε, πρέπει να γίνει καλύτερη γενικά εκτίμηση των συνθήκων. Πολλές φορές ε, είναι μόνο κατόνομα όλα αυτά. Εθνικά δεν μπορούν να υποστηριχθούν τα προγράμματα λόγω των ε, κανόνων κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο και οι συνέργειες αλλά και τα διευθυντικά ταμεία δεν είναι, μάλλον συνέργεια μεταξύ του 2020 και ε, των υπόλοιπων στοιχείων δεν γίνεται ακόμα ακριβώς. Και τέλος σας προσκαλώ όλους στην εκδήλωση που διοργανώνω τη Δευτέρα, όπου και ο ίδιος ο κύριος Σομοέντας, ο Επίτροπος, θα είναι εκεί για να κάνει συγκεκριμένε 10 ε, συστάσεις, ακριβώς για το πώς μπορούμε το πρόγραμμα να το καταστήσουμε πιο φιλικό προς Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ιδέα. Κυρία Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ την Σολεδάδ για το σχέδιο έκθεσής της και σας ευχαριστώ και την Επιτροπή για τη συνεργασία. Συμφωνώ με τους ομιλητές που είπαν ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην πρόταση. Σαφής διάκριση μεταξύ της ε, αμυντικής ε, και πολιτικής έρευνας από την άλλη. Ο θετικός τόνος που δίνεται για τον ορίζοντα 2020, ε, και εγώ συμφωνώ, ε, όμως θα πρέπει να καταστεί πιο σαφή η αξία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Μπορώ να αναφερθώ σε αρκετά στοιχεία, όμω θα ήθελα να, πω, να σταθώ σε αυτά που λείπουν κατά τη γνώμη από την έκθεση ή στα σημεία με τα οποία διαφωνώ. Πρώτον, είναι μάλλον αρνητική η έκθεση ότι αφορά τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο Horizon 2020. Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμη σημασία, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε και να υπερασπιστούμε τα ε, συμφέροντα των επιχειρήσεών μα στο οικοσύστημα τη καινοτομία. Πολύ συχνά πρόκειται και για μικρομεσαίε επιχειρήσει που έτσι μεγαλώνουν υπό την αιγίδα αυτών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία που λάβαμε την Τρίτη το πρωί κατά τη διάρκεια τη ομάδα εργασία ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η προστιθέμενη αξία υπάρχει. Δεύτερον, η έκθεση κάνει ε, μνήα ε, στο κριτήριο της αριστείας και αυτό είναι σημαντικό. Όμως δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι ε, θέλετε να εισαγάγετε την γεωγραφική διασπορά ως υποκριτήριο. Δεν γίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη μου σε καμία περίπτωση. Ορίζον 2020 θα πρέπει να αφορά τη χρηματοδότηση έργων αριστείας και δεν είναι σε καμία περίπτωση τμήμα της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής. Είμαι βέβαια υπέρμαχος ε, της περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με τα διευθυντικά ταμεία. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ένα βαθμό μια πτυχή έρευνα και ανάπτυξη, όμω θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να κλείσουμε το χάσμα μεταξύ των 13 και 15 χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι η EU 13 ε, σχεδόν δεν κάνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό δεν, δεν είναι παράλογο ότι έχουν ε, δρόμο μπροστά τους ε, για να λάβουν και μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το 2020. Για μένα υπάρχει κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο. Ο ΡΙΖΟΝ 2020 ως ε, πρόγραμμα ερευνητικό επιφέρει τεράστια προσθέμενη αξία στην οικοδόμηση γνώσης και συμβάλλει σε μια καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία και θέλω αυτή η ισορροπία μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης αφενός και καινοτομία αφετέρου να διατηρηθεί. Νομίζω ότι τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει ε, να ε, διαδραματίζουν το ρόλο καταλήτη για μια ισχυρή ε, και ανταγωνιστική οικονομία. Προσβλέπω στη συνέχιση τη συνεργασία με τη Σολεδάδη και του άλλου οικειώτε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριο Τελόντεκ, μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω το σχέδιο εκθέσης του εισηγητή. Πιστεύω πως είναι στη σωστή κατεύθυνση για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Ε, νομίζω πως ε, συμφωνούμε με την δομή του προγράμματος. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, ε, αλλά προτείνεται μείωση της γραφειοκρατίας. Έπειτα, η έλλειψη δαπανών σε επίπεδο κρατών μελών είναι πρόβλημα. Είναι μία από τις αιτίε ε, υπερβολικών αιτήσεων ε, χρηματοδότηση από το Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο να τηρήσει τις υποσχέσεις της στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Μετά, η αρχή της αριστείας. Είναι το βασικό κριτήριο που διέπει και τους τρεις πυλώνες. Οι δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών είναι κάτι που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για δημιουργία ικανοτήτων, αλλά ε, ως στόχος πολιτικής. Στόχος είναι να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ζητούμενο στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι πώς θα αξιολογήσουμε ε, τα έργα μας παρουσιάστηκε και στο παρελθόν μια μελέτη που αφορούσε αυτό το θέμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να περικόψει τις δαπάνες για την επιστημονική και περιβαλλοντική έρευνα. Πρέπει να πείσουμε να έρθουν ταλέντα στην Ευρώπη για να εργαστούν στον χώρο αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ω συντονιστής του ΕΛΚ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Λυπάμαι πολύ για την ε, εξέλιξη ε, των ε, εργασιών μας σήμερα, αλλά κάτι δεν πήγε καλά με τους χρόνους ομιλίας. Αυτό να το προσέξουμε σας παρακαλώ. Μετά, έχουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση, έχουμε τους κανόνες, έχουμε τον τους ε, το στο και τον ορίζοντα 2020. Έχουμε δηλαδή στην ουσία συγχωνεύσει τέσσερις εκθέσεις σε μία. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία διαβούλευσης και όταν βρισκόμαστε σε επίπεδο επιτροπής θα έπρεπε ίσως την επόμενη φορά να δώσουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να καταφέρουμε να εξετάσουμε όλες τις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση και, όλες, και την κάθε μία έκθεση ξεχωριστά. Αυτό που έγινε τώρα ε, δεν επιτρέπεται. Και τα ίδια έγιναν και με το FP9. Καταλήγουμε να μην έχουμε χρόνο να πετάμε ακρονίμια και λέξεις χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνουν. Τώρα, ε, επί της ουσίας, ε, θα ήμουν λίγο πιο φιλόδοξος με τον προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος πρότεινε έναν προϋπολογισμό 120 δισεκατομμυρίων. Ε, εγώ δεν θα πρότεινα κάποιον μεγαλύτερο αριθμό, αλλά θα πω τα εξή, ότι μέχρι το 2030 έχουμε πει να αυξήσουμε το μερίδιο του προϋπολογισμού που θα πηγαίνει στην έρευνα και την ανάπτυξη. Με καθαρά και απλά μαθηματικά θα έπρεπε το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο να έχει πολύ μεγαλύτερα κονδύλια. Εάν δεν καταφέρουμε έστω τα μισά από αυτά τα κονδύλια να ε, τα αξιοποιήσουμε και να τα ζητήσουμε από το Συμβούλιο, που έτσι κι έχει αποφασίσει ε, ήδη να ε, τα διαθέσει, τότε δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να ξανασκεφτείτε την πρόταση του Προέδρου για την αύξηση κατά 120 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να δώσουμε τουλάχιστον την εντύπωση ότι κάτι κάνουμε. Μετά, ε, δεν αναφέρθηκαν καθόλου κανόνες συμμετοχή σήμερα και αυτό νομίζω είναι ένα απόσπαστο στο κομμάτι της ενδιαμέσης αναθεώρησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς γιατί ε, θα μας εξηγήσει το τι συμβαίνει με τις υπερβολικές, υπεράριθμες εγγραφές. Πρέπει λοιπόν να διαλευκάνουμε τα, την κατάσταση, να δούμε τι έχει συμβεί εδώ και γιατί. Μετά, ε, θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του, των κανόνων να δούμε πώς θα μειώσουμε τους ελέγχους και πώς θα επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Αυτό έχει να κάνει με την απλοποίηση που έτσι κι αλλιώς έχει ζητήσει η Επιτροπή για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν, να διορτηθούμε αν πραγματικά χρειάζονται τρία επίπεδα ελέγχου. Είμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού και με το Ελεκτικό Συνέδριο έτσι κι αλλιώς σε επαφή και νομίζω πως κάποια, κάποια έλεγχη είναι περιττή. Μετά, συνέργειες. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Η διεύρυνση και η σύνδεση της διεύρυνσης με τα διαρθρωτικά ε, ταμεία. Και πραγματικά νομίζω πως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεταφέρουμε κονδύλια από το ένα ταμείο στο άλλο και να χρησιμοποιήσουμε τις κοινοπραξίες έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες, να δημιουργηθούν πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα δημιουργήσουν μεγάλη μόχλευση έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια. Τέλος, νομίζω πως όταν κάνουμε λόγο για καινοτομία ή όπως το είπε και ο Επίτροπος για, για τη χρήση του ε, ESE, να δούμε τα προβλήματα και να δούμε τι, προσπαθούμε, τι ελλείψεις προσπαθούμε να καλύψουμε με ε, τα κονδύλια. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να εξεταστεί αυτό έτσι ώστε να δημιουργηθούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, οικονομική ανάπτυξη, η ε, αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα, λοιπόν, χρειάζεται αξιολόγηση από όλες τις απόψεις τέλος, κάτι που ήδη ακούστηκε, ε, η εισηγήτρια με βρίσκει αντίθετο σε κάποια πράγματα. 20 χρόνια είμαστε εδώ και κάνουμε τα ίδια πράγματα. Είναι το μοναδικό, ε, η μοναδική εκθέση που αναφέρει την αριστεία. Ε, έχουμε θέματα ισότητας, γεωγραφικά θέματα, αλλά εάν αρχίσουμε να προσθέτουμε κι άλλα, δεν θα έχουμε τέλος. Θα ανοίξουμε το κουτί της πανδώρας, θα εμφανίσουμε χίλια δύο διαφορετικά κριτήρια. Σίγουρα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, να στηρίξουμε τους, ε, τις ε, νέε επιχειρήσεις, να στηρίξουμε το ένα το άλλο, αλλά η αριστεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Διακόπτει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συγγήτρια θα τοποθετηθεί στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, στήριξη στην πρότασή μου να χρηματοδοτήσουμε το FP9. Τώρα, κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι και για προσχάνη συντομία ε, συμφωνώ με το όσα είπαν οι συνάδελφοι του ΕΛΚΑ ε, και να υπογραμμίσω επίσης την εξαιρετική παρέμβαση του συναδέλφου της ΑΛΤΕ, την οποία συνυπογράφω πλήρως. Να κάνω μόνο μια επιλέον παρατήρηση. εκείνο το κομμάτι που αναφέρεται στη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις μεγάλες βιομηχανίες στο πλαίσιο της ε, καινοτομίας και της έρευνας. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πολύ να προσέξουμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο μήνυμα που να είναι ανησυχητικό. Γιατί εγώ προέρχομαι από μια περιοχή της Υπήρου, από μια χώρα όπου η χώρα στο σύνολό της δεν επιφτάνει τους στόχους που θα έπρεπε στην έρευνα. Αλλά η περιφέρεια από την οποία εγώ προέρχομαι, η Νοβαρδία, ε, είναι ένας τομέας που είναι γνωστό σε όλη την Ήπειρο ε, για την έρευνα και τεκμηριώνει ότι η διάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 31 συγκεκριμένα ε, δεν είναι σωστή, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά επίπεδα στήριξης στην έρευνα ανάμεσα στη βιομηχανία και το Πανεπιστήμιο. Είναι επικίνδυνο να μεταφερθεί το σύστημα των grants στα, πανεπιστήμια και των loans στα... Ε, στις επιχειρήσεις. Τα δύο προγράμματα πρέπει να συγκλίνουν γιατί η ισχύ της έρευνας και της καινοτομίας είναι η οικοδόμηση μιας συνεργασίας επίσης ώρες ανάμεσα στο πανεπιστημιακό χώρο και τις μεγάλες εταιρείε. Ε, και ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σε θέση να κάνουν καινοτομία αν, στηριχτούν, αν στηριχτεί και η μεγάλη βιομηχανία το βλέπω στην επικράτειά μου. Ε, αυτό το φαινόμενο σύγκληση ανάμεσα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μεγάλε επιχειρήσει και τα ε, πανεπιστήμια είναι ορατή και απτή. Εάν θεωρήσουμε τη μεγάλη βιομηχανία όρημη και τη αναθέσουμε το έργο τη αυτοχρηματοδότηση τη έρευνα, θα ε, οδηγηθούμε σε μια αποκόλληση που θα σημάνει την ε, μείωση των ήδη χαμηλών επιπέδων έρευνα στην ε, ε, Ήπειρό μα. Στην παράγραφο 31 λοιπόν θα πρέπει να εξισορροπηθεί αυτό το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ο κύριος τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι και Γενικός Διευθυντής. Δύο λεφτά. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο βέβαια, δεν, έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς να, να, συγχαρώ το EPRS για αυτή την έκθεση αξιολόγηση σε πολύ εντυπωσιακή εργασία, αλλά φυσικά πρώτα να συγχαρώ την κυρία Καμπεσόν για τη δική της έκθεση και τους κοιόδης για τα όσα κατάφεραν είναι μια καλή, ένας καλός αντικατοπτρισμός των όσων ισχύουν. Είναι δίκαιη πιστεύω αυτή η έκθεση, αλλά αν μιλάμε για την επιτυχία του Horizon 2020 πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εσείς επιμείνατε για την αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων. 40% των συμμετεχόντων είναι νεοαφιχθέντες. Εσείς μιλήσατε για απλοποίηση, γι' αυτό είναι τόσο προσαρμοσμένο το πρόγραμμα και είναι προσιτό. Ε, επίσης, εσείς ζητήσατε μικρότερο χρονικό διάστημα για την χορήγηση, την ε, πραγματική χορήγηση των χρημάτων. Είμαστε τώρα στους 8 και κάποιες φορές και στους 6 μήνες. Οπότε, από αυτή την άποψη, νομίζω πως η επιτυχία οφείλεται στη δική σας συμβολή και προσπάθεια. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Δεν σημαίνει πως όλα είναι τέλεια βέβαια. Και η έκθεση της κυρίας Καμπεσόν λέει ότι μπορούν να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις. Έχουμε μεγάλη συμβολή και μεγάλα πολλά αιτήματα που μας προέρχονται από διάφορα ενεργητικά κέντρα. Εχθές είχαμε το ε, επέτειο του ERC. Ε, είναι, ε, είναι πραγματικά απίστευτο το ότι καταφέρνουμε στις επιστήμες και στην κοινοτομία. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και η πρότασή σας για 100 δις είναι καλύτερη από τα 80 στα οποία καταλήξαμε τελικά. Αλλά αυτή είναι η βασική μου... Ε, άποψη. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, ε, την διαδικασία σε δύο, ε, αξιολόγηση σε δύο στάδια, βελτιστοποίηση. Υπάρχουν ένα σωρό θετικέ προτάσεις. Υπάρχει ένα στοιχείο όμως στην έκθεση που είναι δύσκολο να το δεχτούμε και αυτό είναι η προσθήκη ενός γεωγραφικού κριτηρίου στην ε, διαδικασία αξιολόγηση. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα αξιολόγηση, αριστείας. Εάν όμως αρχίσουμε να επιλέγουμε τα προγράμματα με γεωγραφικά κριτήρια νομίζω πως θα χάσουμε και πιστεύω πως αυτό δεν θα είναι προς όφελος της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το μόνο πράγμα λοιπόν που έχουμε ζήτημα. Σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε να δούμε περισσότερες ε, περιοχές αριστείας ή ότι δεν θέλουμε να περισσότερες χώρες να ωφεληθούν από το ορίζον 2020. Όχι βέβαια. Γι' αυτό και ακριβώς τονίζουμε τη συνεργασία με τα διευθυντικά ταμεία και συνεργαζόμαστε τόσο ε, σκληρά με τους συναδέλφους της DG Regio γιατί για την ώρα που τα 300 δις έχουν ε, κρατήσει 60 δις για τη δημιουργία δυνατοτήτων για την καινοτομία. Αυτό δεν είναι δουλειά του Horizon 2020, είναι δουλειά των διευθυντικών ταμείων. Το Horizon 2020 θέλει να οθήσει την αριστεία ε, και πρέπει αυτοί οι δύο στόχοι να μείνουν χωριστοί. Ήταν, φανταστική πάντως η συνεργασία και προσβλέπω στη συνεργασία και στο επόμενο διάστημα. Μαζί σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ. Όντως η συνεργασία είναι μακροπρόθεσμη μεταξύ, μεταξύ μας. Έχετε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις. Παρακαλώ μας να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Πολύ χαίρομαι με τις απόψεις. Δεν είναι διευθυντικό ταμείο εδώ αυτό. Υπάρχουν άλλα ταμεία γι' αυτά. Άρα, όσον αφορά ε, ισότητα ε, φύλων, ε, γεωγραφική κατανομή κτλ. Αυτά είναι θέματα των διευθυντικών ταμείων. Εμείς θέλουμε να, εδώ να τονίσουμε την αριστεία. Αυτό είναι ο βασικός και κεντρικός στόχος και είναι δύσκολο να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα. Αυτά. Να σχολιάσω κι εγώ κάτι στη συνέχεια αυτού. Είχαμε μια σχετική έκθεση που ποσοτικοποίησε αυτά που είπατε. Ε, δύο τρίτα των, ε, της βελτίωσης επιδόσεων προέρχονται από ε, την αντιγραφή ήδη άλλων προτάσεων που υπάρχουν. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό της έρευνας και είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία, δηλαδή η αξιολόγηση των γενικών επιδόσεων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε τώρα το λόγο, κυρία Συγκεντριά. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για τα σχόλια και σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω. Να κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις και δύο σχόλια, γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την επίτευξη συνένεση όσον αφορά τη συμμετοχή τη βιομηχανία. Εγώ δεν θέλω να νομίζετε πω δεν θέλω να αποφύγω κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Είπα ότι είναι απαραίτητο για να είναι η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Θα πρέπει όμως να δούμε με ποιο τρόπο θα συμμετέχει καλύτερα, σωστότερα και πώς θα έχουμε, ε, δώσουμε τις περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να βελτιωθούν για το κριτήριο το γεωγραφικό. Ε, ναι, το γνωρίζω ότι αυτό θα άνοιγε τη συζήτηση σχετικά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση για να φτιάξουμε περισσότερα κέντρα αριστείας, περισσότερες περιφέρειες αριστείας. Χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο νέους ερευνητές. Εν πάση περιπτώσει, για να τα πω σύστημα... Ε, Και αυτό είναι ένα project, ένα υπόδειγμα για το πώς οικοδομείται η Ευρώπη. Ε, οικοδομείται με μια ουσιαστική συνένεση και είναι σίγουρο ότι στην εβδομάδα που θα, έχω, ε, θα μας έρθει, που θα έχουμε ακόμα χρόνο για δουλειά, θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Είναι το εγγύς μέλλον αυτό το επόμενο πρόγραμμα και πρέπει να ε, έχουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Okay, okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν σαφείς. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό ε, όποιος από εσάς θέλει κάτι να προσθέσει ή να κάνει μια ερώτηση στους προσκεκλημένους επιστήμονες και στον κύριο Γενικό Διευθυντή. Σας ευχαριστώ πολύ επί τη ευκαιρία που ήσασταν σύντομος. Θα μπορούσατε να προσθέσετε και κάτι αν θέλετε. Ναι. Ένα από τα προβλήματα που συναντήσαμε στην αξιολόγηση είναι το πώς να συνδέσουμε την έρευνα και την αριστεία με τη μείωση ε, των διαφορών ανάμεσα στις περιφέρειες. Νομίζω πως σε γενικές γράμμες γνωρίζουμε τις ε, διάφορες απόψεις που έχουν εκφραστεί. Μία από τις δυνατότητες που δίνουμε στην έκθεση είναι να αυξηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων. Έτσι υπάρχουν οι ερευνητές αριστείας που θα ε, κάνουν το ερευνητικό τους έργο σε ορισμένους τομείς, αλλά να υπάρχει κάποια υποχρέωση να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους και να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους για να αποφεληθούν και η επιστήμονική κοινότητα και οι πολίτες. Αριστεία λοιπόν και ε, διάδοση πληροφοριών για να μειωθούν, τα... να μειωθούν οι διαφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω κάτι στον τελευταίο ομιλητή. Η αύξηση της συμμετοχής είναι λάθος αν γίνει χωρίς σωστή πρώτερη αξιολόγηση των γεωγραφικών ή έμφυλων κριτηρίων. Δεν πρέπει να συγχαίουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Η διεύρυνση της συμμετοχής δεν σημαίνει μείωση της αριστείας, η περιορισμό αυτής με οποιοδήποτε τρόπο το να ψάχνουμε διάφορα μέσα διεύθυνση της ε, συμμετοχής, τότε δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να σταματήσουν να γίνονται αξιολογήσεις προγραμμάτων και έργων. Πάντα πρέπει να ισχύουν τα κριτήρια της αριστείας. Το να δημιουργήσεις όμως κέντρα αριστείας για συγκεκριμένους τομείς, όπως έχει κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπεύει να συνεχίσει να το κάνει και να αυξήσει τα κέντρα στο μέλλον, ε, θα οδηγήσει ταλαντούχους ε, επιστήμονες και από λιγότερο αναπτυγμένες ας πούμε χώρα να ε, δηλώνουν συμμετοχή για επιστημονικά προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά. Συνολικά, έξι χώρες έλαβαν το 68% της χρηματοδότησης από τον ορίζοντα 2020. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, γιατί οι επιστήμονες αυτοί και τα προγράμματα ήταν τα καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να εμποδίσουμε την δυνατότητα δημιουργίας νέων προγραμμάτων που θα προσελκύσουν νέα ταλέντα, ειδικά από αυτές τις χώρες που ε, δεν έχουν την ίδια συμμετοχή, την ίδια επιθετική ας πούμε στάση στις αιτήσει για χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Μόνο μια ερώτηση έχω για την ανοιχτή πρόσβαση. Ε, κάποτε είχαμε συνεισφέρει και εμείς ε, στη δημιουργία ενός ανοιχτού πιλωτικού επιστημονικού προγράμματος. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι έχει γίνει με αυτό το πρόγραμμα, διότι από όσο ξέρω εγώ είχαμε πολλές φιλόδοξες ε, προβλέψεις, όμως είδαμε πολλούς φραγμούς. Υπήρχαν προβλήματα με τη βιομηχανία, προβλήματα με τους εταίρους, ε, ιδιαίτερα όπου υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον. Στα δεδομένα, προσωπικά δεδομένα, είχαμε πρόβλημα και στις ε, υποδομές. Είχαμε αρχίσει μάλιστα να δημιουργούμε ένα επιστημονικό νέφος πληροφοριών. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε ανοιχτό και να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά τότε μάλιστα είχαμε πει ότι πρέπει να είναι ε, όσο ανοιχτό γίνεται. Τι έχει γίνει εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Ναι, λέει ο κύριος Έλλερ, απαντήστε. Είναι όντως ε, πραγματική ερώτηση αυτή που σας έκανα. Ε, να απαντήσω στην κυρία Κοντρίτσκα σε ό,τι αφορά τις ε, δραστηριότητες διεύρυνσης. Στη Λάρνακα, στην Κύπρο είχαμε μια τέτοια εκδήλωση. Εγώ είμαι φίλος αυτών των δράσεων ε, και συμπεριλαμβάνοντας τον ορίζοντα 2020. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όμως γεωγραφικά κριτήρια παντού. Επίσης αυτές οι δραστηριότητες διεύρυνσης ε, εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την αριστεία. Στόχο έχουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Τώρα, για να απαντήσω στον κύριο Έλλερ, καταρχάς υπάρχει γενικότερη προθυμία συμμετοχής ε, στα, στην ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα. Το 60% είναι υπέρ. Όμως πρέπει να το πω και το είπατε κι εσείς ότι υπάρχει ένα opt-out γιατί οι μικρές εταιρείε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να μοιράζονται την δική του πληροφορία, τα δικά του δεδομένα, ακριβώ γιατί είναι, αυτά είναι τα στοιχεία που τους κάνουν ανταγωνιστικού. Το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Υπολογιστικό Νέφος περιέχει δεδομένα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα δεδομένα θα είναι σωστά αποθηκευμένα, θα είναι προσβάσιμα και θα είναι ασφαλή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλό που κάνουμε αυτή την ε, συζήτηση. Και εμείς βέβαια ως Επιτροπή Ήτρε είμαστε αρμόδια για όλο το πρόγραμμα. Η κυρία Καπέθαν Ρουίρ. Μια ερώτηση στο Διευθυντή της Επιτροπής. σε σχέση με την σχέση ε, ΣΔΙΤ. Δεν την αμφισβητώ γιατί είναι απαραίτητη. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στα δημόσια χρήματα που αφιερώνονται στην προώθηση της έρευνας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς ε, στα θέματα, θέματα ας πούμε, υγείας ή φαρμάκων, όπου η δημόσια συμμετοχή είναι απαραίτητη. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι και αυτό ότι το σύνολο του πληθυσμού θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας που συγχρηματοδοτείται από ΣΔΙΤ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Γενικό Διευθυντή, τους επιστήμονές μας, όλους τους συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση που ήταν εξαιρετικά σημαντική. Δεν έχουμε πολλές ε, ευκαιρίες ε, ανταλλαγής απόψεων στην Ήτρα για τόσο σημαντικά θέματα. Λοιπόν, ε, τροπολογίες μέχρι την 31η Μαρτίου, εξέταση των τροπολογιών 24-25 Απριλίου του 2017, και θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο τότε σε σχέση με σήμερα για αυτή τη συζήτηση. Τουλάχιστον 90 λεπτά. Εντάξει, βέβαια σχεδόν μια ώρα τα συζητάμε τώρα εδώ σήμερα, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο για αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πραγματικά κέρια σημασία αρμοδιότητα τη Επιτροπή ε, Ήτρε. Κανεί ε, δεν τη μοιράζεται αυτή την αρμοδιότητα μαζί μα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μα. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τους συμμετέχοντες. Τελευταίο σημείο στη μέση διάταξη, ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ασφάλεια της, ε, του εφοδιασμού φυσικού αερίου. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας δύο λεπτά. Κύριε Έλε. In terms Για την τροπολογία έχω ένα ερώτημα. Θα υπάρξει έκθεση για τους κανόνες ή όχι. Αν όχι, θα πρέπει να διαβρύνουμε τις τροπολογίες για τον ορίζοντα. Αυτά θα δούμε στους συντονιστές στην Επιτροπή Ήτρα, γιατί εμείς είμαστε αποκλειστικά αρμόδιοι. Αν δεν κάνουμε όμως ε, έκθεση για, τη, για τους κανόνες, πρέπει να τροποποιήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με τους κανόνες. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. μάλλον όλα μαζί, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Εξαρτάται από τους συντονιστές, γιατί καθορίζουν τι θα υπάρχει στην έκθεσή μας. Κανονικά ναι και εσωτερικός κανονισμός. Τροπολογίες, παρακαλώ, κυρία Καπεθάνου Ρουίτ, γιατί είστε αρμόδια. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Είναι δύσκολο να έχουμε άλλη έκθεση και είναι απαραίτητη και να έχουμε και χρόνο για να απαντήσει ίσα ίσα ο Γενικός Διευθυντής. Εντάξει, έχουμε όλες τις τροπολογίες για αυτό το θέμα. Τελευταίο. Πολύ σύντομα, λοιπόν, ενημέρωση για τις ε, διαπραγματεύσεις ασφάλεια μυθοδιασμού. Η Ήτρε ε, ενέκρινε στις 13 Οκτωβρίου την εντολή διπραγμάτευσης του Συμβούλου την 1η Φεβρουαρίου Τρέχοντό, σχεδόν 6 μήνες αργότερα δηλαδή. Να πω εν συντομία ότι το Συμβούλιο αποδυνάμωσε την πρότασή μας που ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ξεκάθαρη και είχαμε την ίδια προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιφερειακή προσέγγιση και σημαντικές αναφορές στην αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό φυσικού αερίου και άλλα ζητήματα που άπτονται της ε, κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και τις ε, όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντική συνεργασία μαζί τους, μπορούμε να πούμε ότι μπροστά μας έχουμε κάποιες σημαντικές δυσκολίες. Ιδίως πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα του συντονισμού σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο ξεπερνά το εθνικό, πώς θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια λοιπόν για τα κράτη-μέλη και πώς θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία και πάλι είναι υποσυζήτηση το θέμα της, ε, των κοινοποιήσεων αλληλεγγύη. Όσο Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε αυτή την αίσθηση. Εμείς την έχουμε βέβαια την έννοια της αλληλεγγύης και είναι σημαντικό να μην είναι μόνο θέμα οικονομικό η αλληλεγγύη να υπάρχει όντως ε, η αίσθηση της αλληλεγγύης και αυτή η προσέγγιση μεταξύ των μελών. Πρέπει όμως να πείσουμε και το Συμβούλιο. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αν δεν ε, ολοκληρώσουμε την επόμενη ε, Δευτέρα, τότε 31η Μαρτίου δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε πριν τα τέλη Απριλίου. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η τελευταία, το τελευταίο σημείο. Κυρία Καπιθόν Ρουή, θέλετε να απαντήσετε. Uh, κύριε Γενική Διευθυντά, θέλει να απαντήσετε στην εισηγήτρια. Το σημαντικό είναι η σύνδεση με τον κλάδο, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά τη ε, ΣΔΙΤ. Όμω, ε, η πρόκληση εδώ είναι όντω οι ΣΔΙΤ να παραμείνουν να, συμφέρουσες για τη βιομηχανία, αλλά και να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τη τις κοινωνιακές προκλήσεις. Για παράδειγμα, στα καινοτόμα φάρμακα, οι προτεραιότητες είναι προτεραιότητε του ΠΟΗ, όχι μόνο δηλαδή του ιδιωτικού κλάδου, παρότι πρόκειται για, για ΣΔΙΤ, αντιμικροβιακή αντίσταση και το καθεξής. Αυτό θέλουμε δηλαδή, οι προτεραιότητε, να είναι προτεραιότητες για το γενικό ε, συμφέρον και όχι μόνο για τον ιδιωτικό κλάδο. Βέβαια είναι δύσκολο να εξευρεθεί αυτή η ισορροπία. Και το δεύτερο, ε, δεύτερο παράδειγμα με τον έμπολα, όπου καταφέραμε η βιομηχανία να αναπτύξει εμβόλιο μέσω των ΣΔΙΤ. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη Απριλίου του 2017 θα έχουμε μια επιπρόσθετη συνάντηση της ΙΤΡΕ στο Στρασβούργο το βράδυ στις 7 ή 8,5. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Γιατί ψηφίζουμε για το FC2. Είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσουμε. 3 Απριλίου λοιπόν στο Στρασβούργο, 7 ή 8.30 το βράδυ. Για μισή ώρα ίσως, 40 λεπτά όχι παραπάνω. Δεν είναι πολύ δύσκολη η ψηφοφορία, όμως είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι θα έχουμε αυτή την ε, επιπρόσθετη συνεδρίαση Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είχαμε αυτή τη συζήτηση και αξιοποιήσαμε στο έπακρο το χρόνο μας. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς που είναι μαζί μας από χθες το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Τα λέμε την άλλη φορά λοιπόν στο Στρασβούργο, συνάδελφοι.